Καλημέρα σα. Πρώτο θέμα σήμερα στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση για την έκθεση του κυρίου Αρλάκη. Νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν. Um, be... Πρέπει να σας ενημερώσω ότι θα γίνει και δεύτερη συνεδρίαση, πιθανότατα στις 20 του μηνός. 28 εδώ, όχι στο Στρασβούργο. 28 δεν θα είμαστε στο Στρασβούργο. 28 του μηνός. Ο κύριος Κασουλίδης, που είναι ο βασικός και ηγητής του ΕΛΚ, θέλει να συζητηθεί σήμερα το θέμα αυτό. Ε, υπόλοιπε την άλλη φορά όταν θα τα έχουμε δει. Είναι πάνω από 400 οι τροπολογίες, οπότε σκληρή δουλειά για τον κύριο Αρλάκη ο οποίος θα προσπαθήσει πραγματικά να κάνει κάποιες συμβαστικές απολογίες. Και θα τις συζητήσουμε στις 28 του μηνός. Θα παρακαλούσα τον κύριο Αρλάκη να αρχίσει τη συζήτηση, να πάρει το λόγο για να ξεκινήσει η σημερινή συζήτηση. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. σα ευχαριστώ όλους ε, και τους συνάδελφους που βρίσκονται σήμερα εδώ και ευχαριστώ και όλους τους συνάδελφους που υπέβαλαν τροπολογίες. Αρχικά ε, με ανησύχησε ο μεγάλος αριθμός των τροπολογιών, αλλά αφού τη διάβασα και μελέτησα, θα πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένο, διότι οι περισσότερες από αυτές είναι βελτιώσεις του κυρίου σώματος της έκθεσης. Η δομή της έκθεσης λοιπόν είναι η ίδια με αυτή του σχεδίου και αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο της συζήτησής μας, των συζητήσεων μάλλον που είχαμε ήδη σε αυτήν την Επιτροπή. Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι κατά με το 70% των τροπολογιών είναι απόλυτα αποδεκτές, απόλυτα αποδεκτό και τις, ε, και έχω θετική γνώμη. Δηλαδή έχω κάποιες διαφωνίες για το υπόλοιπο 30%. Να σας εξηγήσω γιατί. και μόνο 15 τροπολογίες από τις 389, δηλαδή 3,8% μόνο του συνόλου των τροπολογιών θα πρέπει να τις απορρίψω ως έχουν τώρα στη διατύπωσή τους. Αλλά θα μπορούσαμε ίσως να τις συζητήσουμε στις συμβιβαστικές ε, και να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και αυτό το 3,8% στο κύριο σώμα της έκθεσης. Νομίζω λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ένας χρόνος δουλειά άξιζε τον κόπο, ήταν πολύ σημαντική δουλειά. Λάβαμε και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης ε, που συμφωνεί με την έκθεσή μας. Διαφωνώ μόνο με το σημείο 9 εκείνης της γνωμοδότησης, μόνο γιατί το, την εποχή που διατυπώθηκε εκείνη η τροπολογία είχαμε μόνο τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές του Αφγανιστάν και άρα αυτό το σημείο θα πρέπει να αναδιατυπωθεί για να ενημερωθεί με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών. Να πω επίσης ότι η φιλοδοξία αυτής της εργασίας είναι να δημιουργήσουμε μια στρατηγική, όχι ένα απλό σχέδιο δράσης, όχι μια απλή προσέγγιση, εγώ έλαβα κάποιες επικρίσεις από την Κομισιόν ότι πραγματικά δεν χρειάζεται στρατηγική για το Αφγανιστάν αφού έχουμε ήδη ένα πρόγραμμα δράσης. Όμως όλες οι ομάδες του Κοινοβουλίου εντόπισαν στις συζητήσεις ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πραγματική στρατηγική και αυτή ήταν άλλωστε η εντολή που μου εδόθη, γι' αυτό και κατέβαλα κάθε την προσπάθεια για να, την, ε, να ανταποκριθώ σε αυτή. Θα βρείτε λοιπόν μια στρατηγική, όχι ένα είδο χριστουγεννιάτικου δέντρου που συχνά βλέπουμε στα προγράμματα δράσης και τις στρατηγικές που δεν είναι ακριβώ στρατηγικές. Καμιά φορά έχουμε στρατηγικές με 10-11 προτεραιότητες. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι στρατηγική. Η πραγματική στρατηγική θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα σαφή αριθμό, σαφή αριθμό, μικρό αριθμό προτεραιότητων και αυτό αυτό προσθέτει στην αξιοπιστία του εγχειρήματο. Γι' αυτό και εστίασα την έκθεση σε τέσσερις μόνο, τέσσερα μόνο κύρια σημεία Ξέρω ότι το Αφγανιστάν είναι φύσκα στα προβλήματα. Ανάλογα με το ποια αγωνία οπτική θα διαλέξει ο καθένας, θα δει και διαφορετικά προβλήματα να αναδύονται, αλλά το Αφγανιστάν είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως όλοι ξέρουμε, καταρχήν λόγω της διεθνούς τρομοκρατία, το γεγονός ότι πήγαμε εκεί με ένοπλε δυνάμει για να καταπολεμήσουμε την παρουσία των ανθρώπων της Αλκάιντα στη χώρα αυτή. Το γεγονός ότι το Αφγανιστάν είναι η πηγή παροχής όπιου σε ολόκληρη ε, την Ευρώπη και στη Ρωσία 99% της ε, παροχής όπιου και ηρωίνης προέρχεται από το Αφγανιστάν και σε εμάς εδώ στην Ευρώπη και στην Ρωσία που είναι επίσης θύμα της, αφρικανικής, ε, της αυγανικής παραγωγής οποίου, όμως από την πλευρά των Αυγανών η μεγάλη προτεραιότητα δεν είναι η τρομοκρατία ούτε το όπιο. Το πρόβλημά τους είναι η φτώχεια. Το Αφγανιστάν είναι μία από τις δύο-τρεις φτωχότερες χώρες του κόσμου, μαζί με τη Σιέρα Λεόνα και κάποιες άλλες αφρικανικές χώρες. Η φτώχεια σκοτώνει στο Αφγανιστάν περισσότερους ανθρώπους από ό,τι οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Εξαρτάται λοιπόν πώς το βλέπει κανείς. Εμείς είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε μεγάλη ευθύνη για την συνέχιση της βοήθειας. Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή στις δικές μας προτεραιότητες, αλλά εγώ προσπάθησα όσο μπορούσα, ώστε να λάβω υπόψη επίσης ποιες είναι οι προτεραιότητες του αφγανικού λαού, που καταρχήν κατά πολέμηση της στόχιας, που όπως είπα είναι το πιο σημαντικό θέμα τώρα και μακροπρόθεσμα για αυτούς και εξάλλου η μείωση της στόχιας παίζει κρίσιμο ρόλο για την επίλυση την μακροχρόνια των αυγανικών προβλημάτων εν γέννη. Παρά όλα αυτά, εγώ επέμεινα στις προτεραιότητες της Ευρώπης. Και γι' αυτό εστίασα σε τέσσερα σημεία. Πρώτον, η ποιότητα του αντικτύπου της διεθνούς βοήθειας Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η ΕΠΑ βασικά, βασικοί είναι οι δωρητές. Υπάρχουν και άλλοι ίσουν σημασία, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι πάντως προέρχεται από αυτούς τους τρεις ε, ε, δωρητές, τις τρεις περιοχές αυτές. Έπειτα, ειρηνευτική πορεία. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά στρατηγική αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λάβει θέση στην ειρηνευτική διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε ευριακή κατάσταση αλλά μετά από την διάσκεψη του Λονδίνου και του Καμπούλ που επέτυχαν να τονίσουν κάτι πολύ σημαντικό για το Αφγανιστάν, ότι δεν υπάρχει δηλαδή στρατιωτική λύση και ότι οι διαπραγματεύσει με ένα τμήμα των Ταλιμπάν θα πρέπει να ξεκινήσει ω ε, τμήμα μια ειρηνευτική διαδικασία. Μετά από αυτό, αυτές τις δύο ε, διασκέψεις έχουμε ένα, μια πολύ σημαντική καμπή στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, εκπαίδευση της αυγανικής ε, αστυνομίας. Και αυτό είναι θέμα κλειδί ώστε να καθορίσουμε τη στιγμή που οι δικές μας δυνάμεις θα αποσυρθούν από τη χώρα αυτή. Η θέση μου δεν θα ήταν πολύ καλή και είναι πως δεν θα ήταν καλό να αποσυρθούμε άμεσα από το Αφγανιστάν γιατί έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία μπήκαμε στο δέκατο έτος παρουσίας στη χώρα συμβάλαμε στην κατάσταση εκεί και δεν μπορούμε εν μία νυχτή να πούμε τώρα τα παρατάμε, φεύγουμε και δεν μας ενδιαφέρει. Το σημαντικό είναι λοιπόν να αφήσουμε πίσω μας μια χώρα που μπορεί να διατηρήσει την ασφάλειά της, ε, η εκπαίδευση της εθνικής της αστυνομίας ώστε να μπορεί να παρέχει ένα μίνιμουμ στάνταρ ε, ασφάλειας στους Αφγανούς πολίτες και εδώ βελτιώθηκε πολύ η αρχική εκδοχή της εκθέσης μέσω των τροπολογιών και το τέλος είναι, η τελευταίο σημείο είναι οι εναλλακτικέ καλλιέργειες στην ε, καλλιέργεια οποίου. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουν επικριθεί όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει στο Αφγανιστάν για το πρόβλημα του οποίου βασικά λυπούμεθα για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμιά απόπειρα για διατύπωση μιας ε, συνεπούς ε, συνεκτικής στρατηγικής ενός πλάνου ώστε να εξαλειφθεί η καλλιέργεια του όποιου σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο. Εγώ έχω δουλέψει πολλά χρόνια στο Αφγανιστάν για αυτό το θέμα. Και γι' αυτό και προσπάθησα εδώ να προτείνω κάποιες ε, συγκεκριμένους τρόπους. Βασική μου πρόταση είναι ότι χρειάζεται μια στρατηγική για την εξάρθρωση, εξάλληψη της ε, καλλιέργειας του οποίου. Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία και ελπίζω πως αυτό θα το εγκρίνουν οι συνάδελφοι για την εκθέση μου. Είδα τις τροπολογίες και βασικά τις δέχομαι. δέχομαι το, δέχονται και εκείνο το πλαίσιο που εγώ έχω προτείνει και γι' αυτό είμαι και ευτυχής για τη συμβολή των συναδέλφων. παρατηρήσεις για την τροπολογία, τις τροπολογίες και την έκθεση. Είναι μια πολύ χρήσιμη ε, κρίσιμη έκθεση, γραμμένη με το συνηθισμένο στυλ που είναι πιο άμεση, ε, είναι πιο κοντά στη γλώσσα των απλών ανθρώπων και επίσης πιο κοντά στα έγγραφα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Εγώ θαυμάζω το Αμερικανικό Κογκρέσο και τον τρόπο με τον οποίο συντάσσουν έγγραφα. Γράφονται όλα με πολύ κατανοητό, σαφή και άμεσο τρόπο, είναι γεμάτα στοιχεία και πολύ απλή γλώσσα χρησιμοποιούν. Οπότε, κάποιο που δεν είναι εξοικειωμένο με αυτού το είδο τη γλώσσα μπορεί να συγχυστεί από το στυλ μου και το γεγονό ότι όπω εμείς λέμε στην Ιταλία λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη και ορισμένες τροπολογίες αυτό το αντικατοπτρίζουν ότι δηλαδή κάπως προσπαθούν να αμβλύνουν ε, τις εκφράσεις ε, που αρχικά εγώ επέλεξα. Δηλαδή την επιλογή που έκανα για να γράψω αυτή την έκθεση με πολύ άμεσο και ευθύ τρόπο. Όμως η έκθεση αυτή είναι επικριτική γιατί μιλά για νέα στρατηγική και μάλιστα στρατηγική εξόδου. Σήμερα η συζήτηση σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα αφορά την έξοδο από το Αφγανιστάν. Πώς θα μπορέσουμε να φύγουμε από τη χώρα, να την αποκαταστήσουμε τη στρατηγική μας παρουσία με, με πολιτική παρουσία και προσέγγιση και ελπίζω πως αυτό θα το εκτιμήσουν οι συνάδελφοι. <clears throat> Να στραφούμε τώρα στις ε, τροπολογίες. Πολλές τροπολογίες ε, βελτιώνουν ε, το περιεχόμενο της έκθεσης. Για να σας δώσω ε, ένα παράδειγμα, αυτό που, με που μιλάει για το δικαστικό σώμα του Αφγανιστάνου. Δεν αρκεί δηλαδή να εκπαιδευτεί μια αστυνομική δύναμη, ένα αστυνομικό σώμα, αλλά πρέπει να εκπαιδεύσουμε και ένα δικαστικό σώμα παράλληλα με την αστυνομία, γιατί διαφορετικά δεν είναι βέβαιο πως ε, το κράτος δικαίου θα διέπει όλη τη διαδικασία και τη λειτουργία της αστυνομίας. Ε, και εκφράζω την πλήρη μου υποστήριξη γι' αυτό, όπως είναι συντεταγμένο. Για το ίδιο θέμα, δεν δέχτηκα μια άλλη τροπολογία που ήταν κάπως υπερβολική. Δεν υποστηρίζω την ε, κατάσταση διεθνών ε, δικαστών ή εισαγγελέων στο Αφγανιστάν που κάναμε στη Βοσνία, στο Κωσυφοπέδιο και αλλού. Το Αφγανιστάν δεν είναι το ίδιο. Ο ποινικό κώδικας είναι διαφορετικός. Πολύ πιο διαφορετικός από αυτό του κοσυφοπηδίου που ξαναγράφτηκε τελείως από αυτόν της Βοσνίας που είναι παρόμοιο με τους ποινικού κώδικες της Ένωσης. Ο ποινικό κώδικας του Αφγανιστάν είναι ένα περίπλοκο σύστημα με πολλά στοιχεία της Αρίας. Και δεν μπορώ να φανταστώ τους διεθνείς δικαστές και εισαγγελείς να εφαρμόζουν το νόμο της Σαρία. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να βασιστούμε στην εκπαίδευση των δικών τους δικαστών που θα στηρίξουν με δικαιοσύνη τη δουλειά της αστυνομίας δίνοντας το χώρο αυτονομίας και κυριαρχίας που χρειάζονται. δεδομένης της μεγάλης απόστασης που χωρίζει το σύστημα, το ποινικό σύστημα εκεί από το δικό μας. Κάποιες τροπολογίες είπα όχι, όχι επειδή είμαι κατά, αλλά επειδή επικαλύπτουν η μια την άλλη ή που ήδη καλύπτονται από κάποια κομμάτια του κειμένου αυτές. Και θα παρουσιάσω στην επόμενη, την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο κάποιες ε, συμβιβαστικές τροπολογίες σε συνεργασία με τους, με τους είμαστε, είμαι ανοιχτό για συνεργασία και είναι <coughs> ε, εύκολο να κάνουμε συμβιβαστικέ και επίση έτσι δεν θα επιβαρύνουμε πολύ το κείμενο. Τώρα, κάποιε άλλε τροπολογίε όμω είπα όχι γιατί στην ουσία έριχναν πολύ νερό στο κρασί του κειμένου και στην ουσία περιόριζαν ή άλλαζαν το νόημα. Τώρα, λόγω του, του θέματος, τα κείμενα αυτά θα πάνε στο τύπο, θα, πάνε, θα διαβαστούν από τον απλό λαό, από το ευρύ κοινό και γι' αυτό δεν χρειάζεται να είναι πολύ περίπλοκα. Όπως σας είπα υπάρχουν 15 τροπολογίες που δεν μπορώ να δεχτώ γιατί είναι κάπως κατά τη ουσία του... και τη κατεύθυνση τη έκθεση. Αλλά όπω σα είπα, είμαι έτοιμο να το συζητήσω με του συντάκτε, ακόμα και αυτέ, και να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια συμβιβαστική. Αυτέ είναι οι τροπολογίε που τονίζουν τα θετικά στοιχεία, όπως αποκαλούνται, τη παρέμβασή μας στο Αφγανιστάν και καταλήγουν ε, ε περιγράφοντας μια ρόδινη εικόνα για τη χώρα. Για παράδειγμα λένε ότι οι περισσότερες μεγάλες πόλεις και οι περισσότερες επαρχίες του Αφγανιστάν δεν αντιμετωπίζουν σήμερα οποιαδήποτε <laughs> θέμα βίας. Μα αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Γιατί εκεί εκείνη τις τροπολογίες που λένε που επενούν τη διεξαγωγή των τελευταίων εκλογών. Είναι ε, ενάντια στις τροπολογίες άλλων ε, συναδέλφων, των περισσότερων συναδέλφων που είναι πολύ επικριτικοί για τις τελευταίες εκλογές στο Αφγανιστάν και επίσης κάποιες τροπολογίες που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών που τονίζουν υπερβολικά κατά την απόψή μου την πρόοδο που έχει δίθεν σημειωθεί σε αυτόν τον τομέα ενώ εγώ και οι περισσότεροι συνάδελφοι πιστεύουμε ότι είναι ένας τομέας όπου έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος και ένας τομέας όπου θα πρέπει να παρέμβουμε ε, για να γίνουν όλα όσα δεν έχουν γίνει στο παρελθόν. Σε μια άλλη τροπολογία γίνεται σύγκριση, με μια πολύ κατάλληλη σύγκριση ανάμεσα στο 76% των ε, θυμάτων ε, των άμαχων πληθυσμού από τους Τάλιμπαν, ενώ λέει είναι μόνο ενώ λέει είναι 84% από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι, συγγνώμη, 24%. Το 24% δίθεν του ΝΑΤΟ, των θυμάτων του ΝΑΤΟ ήταν, λέει, άμαχος πληθυσμός που σκοτώθηκε κατά κάποιο τρόπο όπως ε, σκότωναν και οι Ταλιμπάν. Αυτή είναι μια σύγκριση που δεν στέκει. Και ζήτησα να αποσυρθεί η τροπολογία αυτή. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια βάση μια διεθνή δύναμη που εφαρμόζει τις συνθήκες της Γενέβης τις, και οφείλει να τις εφαρμόζει και από την άλλη πλευρά έναν ε, στρατό που πολλοί που τους νοιάζουν όλες οι συνθήκες της Γενέβης και όλες οι υπόλοιπες. Ναι, κάνουν το ίδιο λέει, αλλά κάνουν περισσότερα. Μα δεν είναι σωστό να λέμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και ζήτησαν να αποσυρθεί αυτή η ε, τροπολογία. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα έχουμε συνεδρίαση στο Στρασβούργο. Μέχρι τα τέλη αυτή εδώ τη εβδομάδα θα πάρετε προτάσει για συμβιβαστικέ τροπολογίε και έπειτα είπε ο Πρόεδρο θα έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία να συζητήσουμε τι τροπολογίε στην ΑΦΕΤ τον Οκτώβριο στι 28 του μηνό με την Full Επιτροπή. Την πλήρη επιτροπή θα έχουμε δηλαδή πολλές ευκαιρίες και σας ευχαριστώ πολύ για την ε, υπομονή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριος Κασουλίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος των περισσότερων μερών του ΕΛΚ που είναι εκτός έδρας, είναι στη Μαδέρα. Γι' αυτό ε, δεν βρίσκονται εδώ. Εσείς μπήκατε λέει. Ε, Κι εγώ θα ήθελα να ήμουν εκεί, αλλά τι να κάνουμε. Ε, επιτρέψτε μου να σας πω καταρχάς ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αρλάκη. Bonjour. Θέλω να ευχαριστήσω, λέω, τον κύριο Αρλάκη για την έκθεσή του. Έχει πολύ μεγάλη πείρα στο Αφγανιστάν, πολύ μεγαλύτερη από τη δική μας και στην έκθεσή του προσπάθησε να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα, από τα τετριμένα και τονίζει ορισμένα σημεία τα οποία θα έπρεπε να ε, είχαν προσεχθεί στο παρελθόν. Για παράδειγμα, εκεί που λέγει ότι η διεθνής τρομοκρατία και τα ναρκωτικά θα πρέπει να συσχετιστούν. Αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντική παραδοχή ε, και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμιστεί. Επίσης κάνει λόγο για τη φτώχεια και η ένδυα είναι βεβαίως ε, η ρίζα ε, του κακού, του διεθνούς φαινομένου της τρομοκρατίας. Και στο Αφγανιστάν γνωρίζουμε ότι καλλιεργείται υπνοφόρος μήκων. Θέλω όμως να τον ευχαριστήσω και για την προθυμία του και την πρόθεση του να βρούμε ε, κοινά σημεία μέσω συμβιβασμών έτσι ώστε να τύχει της ε, μεγαλύτερης δυνατής υποστήριξης και υπερψήφισης η έκθεση. Για μας το Λαϊκό Κόμμα, για την έκθεση και τη διατύπωσή της, ε, το βασικό θα πρέπει να είναι η σημερινή στρατηγική καταπολέμηση ε, των ανταρτών. Όπως ε, αποφασίστηκε πέρσι όταν ανέλαβε γενικός διοικητής ο στρατηγός Μακρίσταλ. Θα επανέλθω σε αυτό. Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει πολλά από τα λάθη, τα σφάλματα του παρελθόντος, τα οποία αναφέρονται και στην έκθεση. Και μερικοί έχουν κάνει και πολλές τροπολογίες σχετικά. Αυτή η στρατηγική λοιπόν καταπολέμησης ε, των ανταρτών λαμβάνει υπόψη ή προβλέπει ότι και ο στρατός και η αστυνομία θα αναλάβουν τις τύχες χώρες το 2014 και η συμμαχία από τον Ιούλιο του 2011 θα πρέπει να σχεδιάζει αποχώρηση. Ε, η καταπολέμηση λοιπόν ε, του Αντάρτικου δεν σημαίνει μόνο μάχες, αλλά απελευθέρωση περιοχών, εξασφάλιση ε, του πληθυσμού ε, καθημερινά, τήρηση της ασφάλειας και συμμετοχή των αμάχων ε, στη κατασκευή ή ανοικοδόμηση των υποδομών. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Για να πετύχει η στρατηγική αυτή, αυτό θα φανεί από τι χώρα θα αφήσει πίσω της. Θα πρέπει να αφήσει μια χώρα που δεν θα ξαναγίνει παράδεισος για ε, τους ε, τρομοκράτες, ούτε τους σκοταδιστές, ούτε τους φονταμενταλιστές του παρελθόντος. Ορισμένοι λέγουν ότι έχει σχεδόν εξαλειφθεί η Αλκάιτα, άρα θα πρέπει να φύγουν οι σύμμαχοι. Δεν συμφωνώ. Το θέμα δεν είναι ότι τους ε, αποκρούσαμε. Το θέμα είναι να μην ξαναγυρίσουν. Η στρατηγική λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ένα σχέδιο δράσης και αναγνωρίζει, όπως σας είπα, τα σφάλματα και τις ελλείψεις των ε, παρελθόντων ετών και της προηγουμένης στρατηγικής. Επίσης αναγνωρίζει ότι από τώρα και στο εξή θα πρέπει να έχει χρόνο η στρατηγική αυτή για να αναπτυχθεί. Οι συμμαχικέ δυνάμεις και οι αφγανικέ δυνάμει δεν μπορούν να κερδίσουν αποκλειστικά και μόνο μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων και οι Ταλιμπάν και οι υπόλοιποι δεν μπορούν επίσης να κερδίσουν του συμμάχους ε, στρατιωτικά. Επαναλαμβάνω, ε, αναγνωρίζονται κάποια σφάλματα του παρελθόντος, όπως οι προηγούμενες τακτικές εστίασης μόνο ε, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δηλαδή έψαχναν τους τρομοκράτες, ε, τους ε, εξουδετέρωναν και ξαναγυρίζαν στα στρατόπεδα στην ασφάλειά τους. Αυτό ήταν σφάλμα. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο άμαχος πληθυσμός και οι απώλειες και πολλές φορές έγιναν συμβόλαια και αναθέσεις εταιρείες μη στρατιωτικές για στρατιωτικά έργα. Ε, πολλά χρήματα δόθηκαν στις υποδομές, παρόλα αυτά δεν καταπολεμήθηκε η καλλιέργεια της παπαρούνας και το όπιο και η ηρωίνη. Από την άλλη, η πλευρά αναγνωρίζει ε, τα επιτεύγματα η εκθέση, αλλά το συνολικό αποτέλεσμα, ο συνολικός απολογισμός είναι απογοητευτικός. Λοιπόν, εάν η έκθεση που εκδοθεί για αυτές τις ελλείψεις και τα σφάλματα του παρελθόντος συνδυάζει ε, τη σημερινή στρατηγική των συμμαχικών δυνάμεων κατά πολέμηση της εξέγερσης Καταλαβαίνουμε ότι και οι επικρίσεις είναι δίκαιες και ε, αποδεκτές. Από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Σαρλάκη θέλει να λάβει υπόψη του αυτά τα σημαντικά στοιχεία και τη σημαντική σύνδεση και τις συμβαστικές τροπολογίες. Πάντως πρέπει να διαφωνήσω κάτι που άκουσα και θα πρέπει να το πω και αυτό. Ίσως να έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μιλούμε εδώ για μια νέα στρατηγική. Στρατηγική υπάρχει. Στρατηγική καταπολέμησης της εξέγερσης. Ε, και θα πρέπει να τη δώσουμε χρόνο για να ε, αποδώσει. Κατά δεύτερο λόγο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για νέα στρατηγική ξεχωριστή από τη στρατηγική των υπολείπων συμμαχικών δυνάμεων. Δεν είμαστε μόνοι μας εκεί και δεν μπορούμε να αποφασίζουμε μόνοι μας. Ενδεχομένως, αντί να χρησιμοποιήσουμε τον όρο στρατηγική, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο πολιτική ή προσέγγιση και αυτό ενδεχομένως να λύνει το θέμα. Για την πολιτική τώρα διαδικασία. Σίγουρα η τελική έκβαση θα είναι πολιτική. Αλλά θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να αφήσουμε το χρόνο στρατηγική να λειτουργήσει ή να αποδώσει. Αν αρχίσουν από τώρα πλήρης ε, ε, διαπραγματεύσεις, θα είναι σε θέση ισχύω η Ταλιμπάν. Ενώ δεν υπάρχει και κυρία αυτή τη στιγμή. Δεν συμφωνούμε ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αποδωσει αν αρχισουν απο τωρα πληρης διαπραγματευσεις θα ειναι σε θεση ισχυωση τα ταλιμπαν ενω δεν υπαρχει και κυρια αυτη τη στιγμη δεν συμφωνουμε οτι αυτη τη στιγμη θα πρεπει να εγκαταλειφθει η χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ο πρόεδρος Καζάη έχει ήδη κάποιες επαφές με τους Ταλιμπάν, αλλά ο Μουλάς Ομάρ έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και διατρανώνει ότι αργά ή γρήγορα εκείνοι θα ε, επικρατήσουν στρατιωτικά. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή εδώ. Όλες οι δυνάμεις που συμμετέχουν στη σύγκρουση θα πρέπει να συμμετάσχουν και στις διαπραγματεύσεις, όποτε γίνουν αυτές. Δεν θα πρέπει να ε, παραμελούμε, ε, να λησμονούμε κάποιους συμμάχου της Βόρειας Συμμαχία και οι διαπραγματεύσεις του Πρόεδρου Καζάη με του Ταλιμπάν δεν θα πρέπει να ε, γίνουν μια υπόθεση ενδοκοινοτική, δηλαδή στο εσωτερικό της κοινότητας των Παστούν και μόνο. Επίσης υπάρχει και ένα θέμα τοπικής και περιφερειακής διοίκησης και κάποιων τοπικών οπλαρχηγών ε, ανταρτών που βρίσκονται ε, στην πλευρά τη λάθος ή των κακών, όχι επειδή είναι τρομοκράτες ή αντάρτες, αλλά επειδή είναι φτωχοί και δεν ξέρουν πού να στραφούν και σε ποιον να απευθυνθούν. Και τώρα ε, ο κύριος Σαρλάκη έχει και μια καινοτόμα προσέγγιση. Θα πρέπει να, δεχτούμε, να παραδεχτούμε κάποια γεγονότα. Το Αμερικανικό Κογκρέσο ε, το ίδιο έχει αναφερθεί για τα τεράστια ποσά που παίρνουν οι ιδιώτες εταιρείε. Και χάνονται χρήματα καθοδό και πηγαίνουν στα χέρια των οπλαρχηγών που πουλούν προστασία. Και λίγα είναι εκείνα τα χρήματα που πηγαίνουν στους θεσμούς του Αφγανιστάν. Πολύ σωστά τα λέει όλα αυτά η έκθεση. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δώσουμε άφηση αμαρτίων στην κεντρική δίκηση του κυρίου Καρσάη σε ό,τι αφορά τη διαφθορά. Χρειάζεται μια επανεξισορρόπηση εδώ ε, της ε, πρότασης, να μην πηγαίνει κατευθείαν η βοήθεια την κεντρική κυβέρνηση του κυρίου Καρζάη. Θα πρέπει να γίνεται η βοήθεια, να δίδεται μάλλον η βοήθεια σε έργα ε, στους, ε, στις διάφορες περιφέρειες. από το 1830 κανένας δεν έχει καταφέρει να φτιάξει μια κεντρική κυβέρνηση στο Αφγανιστάν που να λειτουργεί. Ε, όλα αυτά λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, με οπλαρχηγούς, με φιλάρχους και με τέτοιες νοοτροπίες. Κάθε χρόνο έρχονται στην Επιτροπή μας εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου και εγώ ρωτούσα τα ίδια με τον κύριο Αρλάκη. Πώς είναι δυνατόν να είναι στη χώρα η στρατή μας και να παραμένει η μεγαλύτερη πηγή οποίου το Αφγανιστάν και για την Ευρώπη και για αλλού. Και μάλιστα έτσι χρηματοδοτούν και τους αντάρτες. Ε, στα πρώτα χρόνια και πριν χαρακτεί αυτή η νέα στρατηγική ε, η καταπολέμηση της τροποκρατίας έβαλε στην άκρη, σε δεύτερη μοίρα θέλετε, την καταπολέμηση των εργατικών. Τώρα το έχουν αναγνωρίσει ότι ήταν σφάλμα και διορθώθηκε σημαντικά και χαίρομαι ε, που ο κύριος Αρλάκη κάνει αυτή τη σύνδεση. Θέλω να θέσω κάτι προσωπικό, χωρίς να επιμείνω. Είμαι κατά των αέριων ψεκασμών για να καταστρέφουν οι, καλλιέργειες της παπαρούνας. Το ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί καλλιεργητές που δεν δέχονται εναλλακτικέ καλλιέργειες και μένουν στην παπαρούνα παρά τους ελέγχους της αφγανικής αστυνομίας. Διερωτώ με τι μήνυμα πρέπει να στείλουμε. Ε, να, να, πούμε ε, ότι θα προχωρήσουμε σε τέτοιους, σε, τέτοιους ψεκασμούς, ότι τους εγκρίνουμε ή να το αποσιωπήσουμε τελείως. Επίσης, ε, για τον Αφγανικό στρατό έχει γίνει μεγάλη πρόοδος, Δεν θα πρέπει να αναφέρεται μόνο η αστυνομία αλλά και ο στρατός, γιατί συμμετέχουν ε, σε μικτές ε, δράσεις με τις συμμαχικέ δυνάμεις. Ο Αφγανικός στρατός θα είναι σε θέση να λάβει τον πλήρη έλεγχο της χώρας μέχρι το 2014. Ο κύριος Αλάκη έχει βέβαια το δικαίωμα να μην ασχολείται με αυτό το θέμα και το δέχομαι ως επιλογή. Ε, είδα κάποιες τροπολογίες που προσπαθούν να το εξετάσουν, ορισμένες όμως δεν ανταποκρίνονται ούτε επαναφέρουν την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ αστυνομία και στρατού και δεν είναι ίσως χρήσιμο. Και για την εκπαίδευση τώρα των αστυνομικών πρέπει να πω ότι ο στρατός δεν μπορεί να εκπαιδεύει την αστυνομία. Γι' αυτό ε, οι στρατοί του ΝΑΤΟ εκεί υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να εκπαιδεύουν αστυνομία. Οι ιδιωτικές επίσης αποδείχθηκαν και αποτελεσματικές και ανεπαρκείς. Και θα πρέπει να σταματήσει η ανάθεση αυτής της υπόθεσης σε ιδιωτικές εταιρείες, όχι αμέσως, αλλά ε, μόλις αυτό γίνει δυνατόν. Ε, αναμένονται άλλοι χίλιοι εκπαιδευτέ αστυνομίας και αυτή τη στιγμή αφηχθούν στη χώρα δεν θα χρειάζονται ιδιωτικές εταιρείε. Και επίσης δεν είναι ελαστικό να είναι κριτήριο πρόσληψης ε, η βασική εκπαίδευση. Εκατό χιλιάδες χρειάζονται δημοσίους υπαλλήλους, αστυνομικούς, στρατιωτικούς. Θα πρέπει να είναι και μορφωμένοι. Θα, πού θα τους βρούμε στο Αφγανιστάν τόσους πολλούς. Που, να πούμε κατά προτίμηση. Ε, με βασική ε, μόρφωση εκπαίδευση και μετά θα δούμε κατά πόσο μπορεί αυτό να εφαρμοστεί. Για τα σχόλια του κυρίου Αλάκη νομίζω τα κάλυψα και επίσης σημείωσα πώς να το πω τα πέντε σχόλια του για κάποιες τροπολογίες που δεν δέχεται ή με δυσκολία μπορεί να τις δεχθεί. Με ορισμένε συμφωνώ, για κάποιες άλλες θα πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε. Παρόλο που είπε κάποια πράγματα στα οποία έχει δίκιο. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα να κάνουμε πολύ καλή δουλειά ε, για να βρούμε κοινό έδαφο και να υποστηριχθεί όσο γίνεται ευρύτερα από το Κοινοβούλιο Έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Νόιζερ και θα ήθελα να θυμίσω σε όλου ότι στις 10.30 θα πρέπει να το κλείσουμε το θέμα αυτό γιατί θα έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο κύριος Νόησερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα ως και ηγητής ε, των σοσιαλιστών και δημοκρατών να ευχαριστήσω ειλικρινά τον κύριο Αρλάκη και αυτό δεν είναι έτσι μια απλή φιλοφρόνηση τύπος ευγενία, αλλά ε, δικαιολογείται από την πολύ μεγάλη εμπειρία και πραγματογνωμοσύνη με την οποία έχει κάνει την έκθεση του κύριο Σαλάκη. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι η δική μας ομάδα κατάφερε να τον πείσει για τις περισσότερες τροπολογίες της και τα επιχειρήματά της και χαίρομαι γι' αυτό. Είμαστε πάντα πρόθυμοι να συζητάμε με ειλικρίνεια ε, οι μικροδιαφορές που παραμένουν νομίζω μπορούν να γεφυρωθούν εύκολα. Είχα διατελέσει και σκιώδης ηγητή στην ε, Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας και πιστεύω ότι και εκείνες οι τροπολογίες ε, έχουν συμπεριληφθεί όλες καλώς στην έκθεσή του. Ένα σημείο μόνο χρειάζεται ενημέρωση. Τώρα, αν έχουμε νέα στρατηγική, νέα πολιτική για το Αφγανιστάν, δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο αλλά δεν είναι πρόγραμμα δράσης. Η έκθεση αυτή ε, αφορά κάτι παραπάνω. Συμφωνούμε με το γενικό προσανατολισμό της έκθεσης, διότι εξετάζει με πάρα πολύ κριτικό μάτι την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Δεν την περιγράφει καθόλου ρόδινα. Είναι μια έκθεση ισόρροπη που λαμβάνει όμως υπόψη και τα θετικά, χωρίς να ευρωποιεί την κατάσταση. Κάτι άλλο που ωφελεί την έκθεση επίσης και είναι και χρήσιμο είναι ότι δεν στρέφεται στο παρελθόν, αλλά στρέφεται στο μέλλον. Δηλαδή δεν θέλει τώρα να αποδώσει ευθύνε και ενοχέ. Είναι στραμμένη προ το μέλλον για να μπορούμε να κάνουμε και μια καλή συζήτηση για το μέλλον. Για μα επίση αποφασιστικό είναι ότι ο προσανατολισμό είναι ευρωπαϊκό, τη Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, και επικεντρώνεται στα καθήκοντα ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε αρμόδιοι γι' αυτό και για να το τονίσω δεν είμαστε η κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ εδώ, είμαστε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ωστόσο, αυτά που κάνει το ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και με ρεαλισμό γιατί τελικά τον αποφασιστικό ρόλο στο Αφγανιστάν το ΝΑΤΟ το διαδραματίζει. Είπα προηγουμένως ότι είναι ρεαλιστική η εκτίμηση της έκθεσης, αλλά Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ε, επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό. Και αυτό είναι σημαντικό να το δούμε και καλύτερο γιατί χρειαζόμαστε μια στρατηγική και μετά το 2014, μετά την ημερομηνία της ε, πλήρους απόσυρσης. Εδώ με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η καταπολέμηση της ένδειας που είχε αρχίσει πριν το 2001 στο Αφγανιστάν και τώρα θα πρέπει να ενταθεί και μετά το 2014 όλος ιδιαίτερος. Γι' αυτό οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν μεγάλο ρόλο και το τονίζω, έχουν μακρά, μακροχρόνια πείρα στο Αφγανιστάν και πάντα θα πρέπει να βασιζόμαστε στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και κινδυνεύει το προσωπικό τους εκεί, όπως και οι ε, δικοί μας στρατιώτες που εμείς τους έχουμε στείλει εκεί με δική μας εντολή. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις επίσης ε, ασχολούνται ιδιαίτερα με την κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί να έχει βελτιωθεί αλλά σε καμία περίπτωση ε, έτσι όπως μας το παρουσιάζουν συχνά. Επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε να οικοδομηθεί η κοινωνία των πολιτών ε, και η στρατηγική ε, που θα συμπεριλαμβάνει και θα ενισχύει τις τοπικές αρχές. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν παράλληλα ε, προωθήσουμε και τονώσουμε την κυριαρχία του κράτους δικαίου εκεί. Υπάρχει εδώ μια προϋπόθεση όμως. Καλύτερη εκπαίδευση της αστυνομίας που θα πρέπει να οργανώσουμε εμείς για να δεύουν και τα δύο αυτά παράλληλα. Μια τελευταία μόνο παρατήρηση για τη διαδικασία συμφιλίωσης που συμπεριλαμβάνει ρητά και τους Ταλιμπάν. Ε, θα πρέπει ε, να κάνουμε μία διαφοροποίηση πάντα. Γιατί μπορεί να έχουμε καμιά δεκαριά ομάδες Ταλιμπάν. Έτσι. Ε, υπάρχουν κάποιοι που είναι τελείως εκτός κάθε συνεργασίας ε, και πρέπει να τους καταπολεμούμε. Είναι όμως κάποιοι άλλοι Ταλιμπάν επίσης ε, που τους πίεσαν για να γίνουν Ταλιμπάν, τους εκβίασαν για να γίνουν Ταλιμπάν για λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς και κατέληξαν εκεί. Σε αυτούς θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να εστιάσουμε την προσοχή μας. Αν θέλουμε όμως να αρχίσουμε μια διαδικασία συμφιλίωσης, αυτή γίνεται μόνο ε, συμπεριλαμβανομένων των Ταλιμπάν. Ευχαριστώ λοιπόν τελειώνοντα και πάλι τον εισηγητή για την κατεύθυνση που παίρνει, για τον προσανατολισμό του, γιατί ανταποκρίνεται και στι δικέ μα ιδέε, και ελπίζω και την άλλη εβδομάδα να συνεχίσουμε την καλή μα συνεργασία και τέλειο Οκτωβρίου, έτσι ώστε στο Κοινοβούλιο να έχουμε μεγάλη υποστήριξη και πλειοψηφία για την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Σόλτ. Äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ γερμανικά θα μιλήσω. Ε, καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του, εισηγητού, του σιώδη εισηγητού της ομάδας μου και των συναδέλφων που είναι και αυτοί σε ημερίδες μελέτη στο εξωτερικό. Εμείς υποστηρίζουμε την προσέγγιση του εισηγητού και την αφετηρία του και θέλουμε να τον, βοηθήσουμε, να τον ευχαριστήσουμε συγγνώμη, και για την προσέγγιση αυτή, αλλά και για την προσπάθεια που κάνει επαναπροσδιορισμού, επανακαθορισμού της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν και τη ε, κοινότητα τη διεθνή από πλευράς ε, των διαφόρων εξελίξεων και ασφαλείας και πολιτικών και οικονομικών και κοινωνικών. Έχει τονιστεί εδώ. Κατά την άποψή μας η έκθεση αποδίδει πολύ καλά την εικόνα του πώς αντιλαμβάνεται ε, ο κόσμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη σύγκρουση εκεί στο Αφγανιστάν και πώς μπορεί να οδηγήσει η γνώμη του ευρωπαϊκού πληθυσμού σε μια νέα πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Αφγανιστάν. Όλοι γνωρίζουμε ότι η στρατιωτική λύση και η συμμετοχή ε, ευρωπαϊκών ε, στρατών και στρατών ε, των χωρών του ΝΑΤΟ είναι κάτι που ο πληθυσμός απορρίπτει. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια απόκληση. Άλλο κάνουν οι κυβερνήσεις και άλλη αίσθηση έχει ο πληθυσμός ή άλλη ε, αντίληψη έχει ο, ο πληθυσμός στην Ευρώπη για το πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η κατάσταση και να αντιμετωπιστεί στο Αφγανιστάν. Πρέπει να καλυφθεί λοιπόν, να κλείσει αυτή η ψαλίδα. Είναι τέσσερις οι μεγάλοι τομείς που θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να ακολουθήσουμε μια νέα πρόπτικη. Και συμφωνούμε και εμείς με αυτούς. Προσωπικά συμφωνώ με τον εισηγητή, το είπε και σήμερα, ότι η λύση δεν είναι στρατιωτική. Ωραία. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει η Ευρώπη να συμμετέχει στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. Πώς θα προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια μη στρατιωτική λύση. γιατί είναι πάρα πολύ περίπλοκα τα προβλήματα στη χώρα και πάρα πολύ βαθιά ριζωμένα. Συμφωνώ επίσης ε, για την ανοικοδόμηση και της δικαιοσύνης και όλων των δομών και των υποδομών και των κεντρικών και των περιφερειακών. Πρόσφατα στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου συζήτησα με Ινδούς συναδέλφους που είπαν ότι έχουν μαζική εκεί παρουσία και με νομικούς για να συζητήσουν ε, ας πούμε το δίκαιο του ανταγωνισμού και άλλα τέτοια σημαντικά ζητήματα οικονομικής φύσεως για να δώσουν νέα εργαλεία και σε εκείνους που ασχολούνται με την οικονομική ζωή του τόπου. Θα πρέπει να τη σκεφτούμε και αυτή την κατάσταση και στις συμβαστικές τροπολογίες μήπως θα μπορούσαμε να τις ενισχύσουμε τις προτάσεις αυτές. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των γυναικών δεν μπορώ να, παρά να συμφωνήσω με τις προαλήσαντες δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών. Το αντίθετο μάλιστα. Ακούμε ότι έχει επιδεινωθεί. Είναι πάρα πολύ επισφαλής και αβέβαιη. Κάτι άλλο που ίσως να μην έχει κυριαρχήσει στη συζήτηση αλλά και στην ανασχόλησή μας ε, με το θέμα αυτό στο μέλλον, όχι μόνο εδώ αλλά και σε άλλες ε, επιτροπές και θα πρέπει να τα ξαναδούμε, είναι τι γίνεται με την παραγωγή ενέργειας εκεί. Δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό για την ε, ε, οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας, για να συμμετέχουν δημοκρατικά οι άνθρωποι στη διαμόρφωση ε, της ζωής τους, της ίδιας και των συνθηκών διαβίωσης. Για να δούμε πώς μπορεί να αναπτυχθεί οικονομικά ε, η χώρα και από ένα άλλο πρίσμα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω πάρα πολύ, αλλά ε, πιστεύω κι εγώ ότι ε, αυτά που έγραψαν οι Financial Times Deutschland για τις εκλογές της 20 ε, Σεπτεμβρίου είναι σωστή. Δεν είναι μόνο σε τέλμα η διαδικασία εκδημοκρατισμού της χώρας, αλλά σε οπισθοδρόμηση. Γιατί εκτός από το θέμα της ασφάλειας, ε, η χαμηλή συμμετοχή σε εκλογές ε, εξηγείται και από ένα δεύτερο στοιχείο που είναι η νοθεία στις εκλογές. Βεβαίως χρειάζεται νέα πολιτική, νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ειλικρινή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μη στρατιωτική, άρα απόσυρση των στρατευμάτων και υποβοήθηση της εσωτερικής διαδικασίας ειρήνευσης της χώρας. Ευχαριστώ. Now, Mrs. please. Ευχαριστώ. Κυρία Κοπά, παρακαλώ. Thank you, Mr. Ε, θα ήθελα να εκφράσω αρχικά τα συγχαρητήριά μου στον συνάδελφο Αρλάκη για την έκθεσή του και να συμφωνήσω επί της αρχής με την προσέγγιση του και τη σκέψη του να πούμε ορισμένα πράγματα με το όνομά τους, με τρόπο που να είναι κατανοητά ε, από τους Ευρωπαίους πολίτες. Εννιά χρόνια παρουσία στο Αφγανιστάν καθιστούν πλέον ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση. Σωστά λοιπόν τονίζεται στην έκθεση ότι τα χρήματα που ξοδεύονται σήμερα σε πολεμικό υλικό θα ήταν πιο λογικό να διοχετεύονται για την εξάλληψη της φτώχειας στη χώρα. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι έχουμε και εμείς ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση και δεν μπορούμε απλώς να την εγκαταλείψουμε στη μοίρα της. Έτσι, η ενδεχόμενη αποχώρηση των δυνάμεων πρέπει να, να γίνει συντονισμένα και σταδιακά, στο πλαίσιο πάντα μια πολιτική λύση που θα εξασφαλίσουμε για το Αφγανιστάν. Η έκθεση που μελετάμε σήμερα και οι τροπολογίες που κατατέθηκαν, ιδιαίτερα σε σχέση με την παράγραφο 32 και 33, αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για να μιλήσουμε για αυτή την πολιτική λύση την οποία προσπαθούμε να σχεδιάσουμε. Αυτή η λύση πρέπει να έχει συγκεκριμένα μέτρα και όχι γενικόλογες ευχές για την εκρίζωση της φτώχειας του Αφγανιστάν. Πρέπει από τώρα να είναι σαφές ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αποκλείσουμε οποιαδήποτε πολιτική δύναμη επιθυμεί το συμβιβασμό και την ειρήνη και πιθανότατα πρέπει να υπάρξει εκτεταμένη αποκέντρωση. Ο στόχος μας πρέπει να είναι μια λύση που θα εμπλέκει την κοινωνία των πολιτών στο Αφγανιστάν και όλες τις μέχρι σήμερα περιθωριοποιημένες ομάδες στις διαδικασίες ειρήνευσης, με ιδιαίτερη προσοχή για τους Παστούν, που πρέπει να αναφέρονται κατά τη γνώμη μου στο κείμενο, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σημερινή εξέγερση και αναπόφευκτα θα αποτελέσουν α, μέρος οποιασδήποτε μελλοντικής πολιτικής λύσης. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί λογοδοσία που είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να καταπολεμηθεί η διαφθορά, την οποία όλοι αναγνωρίζουμε σε κρατικό επίπεδο. Πρέπει επίσης να δούμε το ευρύτερο περιφερειακό περιβάλλον και να σκεφτούμε πού μπορεί να εντοπιστούν κοινά υποφελείς τομεί περιφερειακής συνεργασίας. Με τον σκιώδη εισηγητή της ομάδας μου, ε, τον Νόρμπερ Νέουζερ, προτείνω να τονίσουμε τη σημασία πρωτοβουλειών στον τομέα της διαχείρισης υδάτων, ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ του Αφγανιστάν και των γειτόνων του. Θυμίζω με αυτή την ευκαιρία τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στο Πακιστάν, στη σχέση με τις οποίες πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους πλημμυροπαθείς Αφγανούς πρόσφυγες, αλλά και να αντιμετωπίσουμε πιο σφαιρικά το ζήτημα, αναλύοντας ενδεχομένως καλύτερα τις όποιες πολιτικοστρατηγικές συνέπειες. Κλείνοντας, θέλω να προσθέσω ότι προσωπικά δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με εκείνες τις τροπολογίες που εκφράζουν απογοήτευση για τις πρόσφατες εκλογές, που παρά την προσπάθεια πολλών διεθνών ε, παραγόντων να τις ωρεοποιήσουν, αποτέλεσαν για όλους μας ένα déjà με πρωταγωνιστές τη βία και την οθεία. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σβόμποτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ την έκθεση αυτή πραγματικά καινοτόμα, αλλά και θαραλέα, γιατί θέτει νέα κέντρα βάρους. Δεν ξέρω αν πρόκειται για νέα στρατηγική για συνέχιση της παλιάς. Ο καθένας μπορεί αυτό να το εκτιμήσει διαφορετικά αν πρόκειται για το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πλευράς ΝΑΤΟ είναι σίγουρα νέα στρατηγική. 8-9 χρόνια μετά την έναρξη αυτής της επιχείρησης άρχισε να σκέφτεται το ΝΑΤΟ τι θέλει να πετύχει αλλά και τι μπορεί να πετύχει. Και αν θέλετε ε, να κάνουμε μια σύγκριση των δύο επιχειρήσεων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, έχει κλονιστεί η αντίληψη που λέει επεμβαίνει σε μια χώρα, ρίχνεις μια κυβέρνηση και φέρνεις τη σωτηρία της και αλλάζει το σύμπαν. Αυτό έχει κλονιστεί ως αντίληψη. Έτσι κι αλλιώς εμείς δεν μπορούμε να ε, σώσουμε τον κόσμο και σίγουρα δεν μπορούμε να το κάνουμε με στρατιωτικές επεμβάσεις και με εισβολές, χωρίς να έχει σχεδιαστεί η επόμενη μέρα. Το τι μέλη γενέστε ε, ε, μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων και απεδείχθη σφάλμα αυτό που είπε και λαθασμένο ο πρόεδρος Μπούς ε, αποστολή εξετελέστη. Mission accomplished, το θυμάστε. Και τα αντίστοιχα ισχύουν για το Αφγανιστάν. Οι συζητήσεις τώρα γίνονται συνομιλίες με τους Ταλιμπάν. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά δεν θα πρέπει μετά από 10-12 χρόνια εμείς να αποσυρθούμε και τελικά να έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό να ε, ε, υπάρχει το ίδιο καθεστώς και το ίδιο status quo. Το λέει και η έκθεση αυτό, προσπάθησα να το διευκρινίσω ακόμα περισσότερο σε μία ε, τροπολογία, με ποιους Ταλιμπάν θέλουμε να μιλάμε. Ο συνάδελφος Νόισερ είπε ότι υπάρχουν πολλές ομάδες Ταλιμπάν. Ορισμένοι ε, ονειρεύονται επαναφορά του προηγμένου καθεστώτος για να υποδέχονται μεταξύ άλλων και τρομοκράτες. Αυτό θα πρέπει στη θυσία και με κάθε δύναμη να αποτραπεί, διότι αυτό ήταν στη ρίζα της επέμβασης. Μετά ακούστηκαν διάφορα ευκολόγια. Βεβαίω δεν θέλουμε οι γυναίκε να φοράνε μπουρκα, θέλουμε τα κορίτσια να πηγαίνουν σχολείο. Το θέμα είναι πώ θα το επιβάλλουμε αυτό. Υπάρχουν όρια. Ίσως η έκθεση θα πρέπει να είναι πιο μετριοπαθή ακόμα και αν αυτό είναι κάτι που μα λυπεί. Αλλά να είμαστε ρεαλιστέ, τι μπορούμε να επιβάλλουμε. Λοιπόν, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συζητήσουμε ε, με κάποιε ομάδε τα Λιμπάν. Βέβαια, ο Καρζάη το κάνει ήδη, δεν ξέρω αν είναι σωστό και τι επιπτώσει θα έχει αυτό, αλλά να συνεννοηθούμε με εκείνε τι ομάδε που είναι πρόθυμε, βεβαίω με τη συμμετοχή του στην εξουσία, να εφαρμόσουν κάποιε αρχέ τη δημοκρατία της ισότητας και τα λοιπά και να τις αναγνωρίσουν. Μην νομίζετε ότι θα είναι η ίδια δημοκρατία με εμά, ε, ούτε η ίδια ισότητα που επικρατεί στις δικές μας χώρες. Αλλά ένα ελάχιστο δικαιωμάτων και η διασφάλισή τους είναι απολύτως σωστό. Αυτά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Τα είπαν οι άλλοι συνάδελφοι. Απλώς το δίδαγμα και θα άρχισε να κάνουμε μια Εκθεσία επί της αρχής είναι όχι στη στρατιωτική επέμβαση χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων σχεδιασμός πολιτικός, μη στρατιωτικός δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να είναι απαραίτητη η στρατιωτική επέμβαση για ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, δεν ξέρω ποιος, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πολύ καλύτερα από την αρχή ε, να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα, κάποια διδάγματα. Τι καταλάβαμε από το Ιράκ και από το Αφγανιστάν. Έχουμε βγάλει κάποια ε, συμπεράσματα, έχουμε αποκομίσει μαθήματα, διδάγματα ε, και ε, τακτική για το μέλλον. Η έκθεση αυτή είναι σημαντικό, ουσιαστικό στοιχείο αυτών των διδαγμάτων. Να μην είμαστε αφελείς ότι δεν θα υπάρξει ποτέ πια στρατιωτική επέμβαση πουθενά, αλλά ποτέ πια στρατιωτική επέμβαση χωρίς σαφή πολιτικό σχεδιασμό. Πάντα βεβαίω προσαρμοσμένο στην εκάστοτε χώρα, όχι κανένα γενικό αφηρημένο μοντέλο. Γιατί το Ιράκ και το Αφγανιστάν ήδη από μόνα τους είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε τις ειδικέ καταστάσεις στην κάθε χώρα, γιατί αυτό είναι ολέθριο σφάλμα. Κατά τα άλλα, υπόθηκε ήδη ότι η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή και βάση και μόνο για προβληματισμό και συζήτηση το τι θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον σε παρόμοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάλερ παρακαλώ και να σκέφτεστε και την ώρα σας παρακαλώ πολύ. Ένα τέταρτο έχουμε μόνο. 20 λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην γίνω Φιντέλ Κάστρο. Πολλοί συνάδελφοι είπαν πράγματα με τα οποία σύμφωνο, διότι αυτό μου επιτρέπει να είμαι και πιο σύντομος. Σύμφωνο και εγώ στον ευχαριστήσω τον κύριο Αρλακή, ο οποίος έχει κάνει μια τεράστια δουλειά. Και ε, πολλοί συνάδελφοι το θύμισαν ότι δεν πρέπει να χάνουμε το σύνολο και να χαθούμε μέσα στις λεπτομέρειες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιος είναι ο στρατηγικός μας στόχος αυτή τη χώρα, δηλαδή να βοηθήσουμε την πολιτική διαδικασία να εξελιχθεί στο Αφγανιστάν που θα, θα σημαδέψει και το τέλος της στρατιωτικής κατοχής. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε μια σωστή πολιτική εξέλιξη. Έχουμε τον Καρζάη στην κορυφή και μια πυραμιδοειδή διάρθρωση της εξουσίας αλλά αυτό δεν είναι η αφγανική παράδοση ποτέ δεν λειτουργήσε έτσι το Αφγανιστάν οι Αφγανοί έχουν ένα ε, μοντέλο αποκεντρωμένης δημοκρατίας ή αν θέλετε μία μεικτή κυριαρχία με διάφορα επίπεδα εξουσίας στη χώρα για παράδειγμα στο φορολογικό επίπεδο, στο στρατιωτικό επίπεδο κλπ. Δεν θέλω όμως να, να, να επισέλθω σε άλλες λεπτομέρειες. Υποστηρίζω το κομμάτι εκείνο του ψηφίσματος όπου αποφασίσαμε να επενδύσουμε παραπάνω χρήματα σε αυτήν την πολιτική διαδικασία για την εθνική συμφιλίωση των Αφγανών. Σύμφωνο με τους συναδέλφους, πρόκειται για πολύ απλά πράγματα. Χρειάζεται να έχουμε συνέστηση μια συνέστηση των ιδίων των Αφγανών και μια δέσμευση των Αφγανών ούτως ώστε να ξοπετάξουν την Αλκάιδα από τη χώρα. Χρειαζόμαστε ένα μήνυμο εγγυημένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στο ψήφισμα θα πρέπει λοιπόν εμείς να επικεντρωθούμε σε αυτήν την πολιτική διαδικασία η οποία θα πρέπει να συνοδεύει το Αφγανιστάν για το μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Νέσκι. Θα μιλήσω βουλγαρικά. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Αρλάκη, για την ανάλυση που κάνει. Με πάρα πολύ άμεσο τρόπο και ευθύ. Είναι γεγονός ότι χρειάζεται τέτοιου είδους ανάλυση ε, όταν θέλουμε να προτείνουμε μια νέα προσέγγιση. Μέχρι τώρα η προσέγγιση ήταν μάλλον γενική και αόριστη. Τώρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις λεπτομέρειες και να καταλάβουμε, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να δούμε τι κάναμε λάθος. Έχει δίκιο ο εισηγητής όταν λέει ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα στη δικαιοσύνη, την ασφάλεια, την καταπολέμηση της παραγωγής ε, οποίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή την νευτική και ο γενικός πληθυσμός. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που δεν έχει ζήσει βέβαια τέτοιου είδους προβλήματα, αλλά είχαμε στο παρελθόν άλλα προβλήματα. Είχαμε ένα κράτος το οποίο κατέρευσε και καταλαβαίνω και γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να οικοδομηθούν οι θεσμοί, να υποστηριχθεί η ε, ανάπτυξη, η εκπαίδευση και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή να συμμετέχει ο γενικότερος πληθυσμό στην προσπάθεια αυτή. Για να βγει από τη φτώχεια και να αρχίσει να εργάζεται ο κόσμος και να αρχίσει να δρέπει και τους καρπούς και τα ωφέλη από τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας. Επίσης θα πρέπει να επικεντρωθούμε και ε, στους ηγέτες εκείνους που είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν στην ευτική διαδικασία και να μας βοηθήσουν να αντικρούσουμε τους Ταλιμπάν και να τους αποκρούσουμε. Είναι ο μόνος τρόπος επίτευξης ειρήνης. Είναι λοιπόν πιστεύω πολύ καλό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση αυτή η έκθεση και συγχαίρω τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Από την Επιτροπή, ο κύριος Πολ Τέραν από την ε, Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήθελα απλά να πω από πλευρά τη Κομισιόν ότι προφανώ εργαζόμαστε σε αυτή την έκθεση γιατί είναι μια εξαιρετική ανάλυση, πολύ κέρια ανάλυση των προβλημάτων. Εμείς θελήσαμε να προσέξουμε το γεγονός ότι δεν θέλουμε τώρα να πιαστούμε σε μια, σε μια συζήτηση ε, σημασιολογική για το αν είναι στρατηγική, η νέα προσέγγιση. Το Αφγανιστάν έχει διάφορε στρατηγικέ, εθνική πολιτική στρατηγική, ε, μάλλον στρατηγική για την αντιμετώπιση της στόχης. Η ISAF ασχολείται με το θέμα της ασφάλειας και η αφγανική κυβέρνηση μετά από τη διάσκεψη της Καμπούλ πριν από το καλοκαίρι πρότεινε νέα διοργάνωση σε σύνολα όπου οι δωρητές έχουν συμφωνήσει. Έχει γίνει, έχουν υπάρξει πολλές εξελίξεις. Η κοινότητα των δωρητών θέλει να συνεργαστεί με τους Αφγανούς και να τους βοηθήσει να ε, στερεοποιήσουν τη δομή που έχει ήδη δημιουργηθεί. Και επίσης αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι και κρίσιμο είναι να ελέγξουμε πραγματικά για το τι ποσά συζητάμε όταν λέμε για νέα στρατηγική της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται τα συστήματα και μιλάμε για 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πέντε φορές λιγότερο από αυτό που δίνει η Ιαπωνία το χρόνο. Εάν συγκεντρώσουμε το σύνολο του κοινοτικού προπολογισμού, δηλαδή των, ε, των ε, Είμαστε κάτω από το 1 δις ε, το χρόνο αν προσθέσουμε και τα όσα δίνουν διμερώς στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Και ακόμα λιγότερα, ε, εξακολουθούμε να είμαστε κάτω από αυτά που δίνει η Ιαπωνία και η ΕΠΑ. Δηλαδή, λέμε για νέα στρατηγική, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας γιατί χρήματα μιλάμε, τι ποσά μιλάμε. Γιατί από τη στιγμή που πάει το, η Κομισιόν για έγκριση των προπολογισμών στα κράτη-μέλη και για το Κοινοβούλιο, κράτη-μέλη έχουν και τη δική τους διμερή βοήθεια, επί της οποίας το Κοινοβούλιο δεν έχει έλεγχο. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε υπόψη μας τι, τι, λέμε όταν μιλάμε για νέα στρατηγική νέα προσέγγιση. Κάτι ακόμα. Δεν είμαστε κατά των ιδεών που έχουν προταθεί εδώ, αλλά πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια καλή χαρτογράφηση του τι κάνει η διεθνής κοινότητα στο Αφγανιστάν, ιδιαίτερα τους τελευταίους έξι μήνες, όπου έχουμε εστιάσει την προσοχή όχι μόνο στο τομέα της ασφάλειας, αλλά και στο τομέα της ανάπτυξης και οι Αφγανοί έχουν ε, στην ουσία τοποθετηθεί στην ηγεσία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο μια στρατιωτική απόσυρση, προφανώς συμβαίνει αυτό. και με τις διαδοχικές συνεδριάσεις του ΝΑΤΟ λοιπά, Αλλά και πολιτική απόσυρση, δηλαδή προσπαθούμε να πιάσουμε πια τις πίσω θέσεις τα όσα γίνονται εκεί, ακόμα και σε επίπεδο πολιτικών ενεργειών και δράσεων. Στην ουσία τα όσα έγιναν εκεί παγιώθηκαν το τελευταίο χρόνο ε, και ε, συμφωνούμε 100% με την έγκυρη ανάλυση που γίνεται όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, γενικότερα στο Αφγανιστάν και την ανικανότητα στην οποία, την οποία διαπιστώνει η διεθνή κοινότητα δεν μπορεί να, δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να σας πω κάτι ακόμα Η εθνική κυβέρνηση στην ουσία προτείνεται ως ε, ο τρόπος για να λυθεί το θέμα και προτάθηκε επίσης ότι το Αφγανιστάν ανέκαθεν ήταν αποκεντρωμένο κράτος και πρέπει και πάλι να αποκεντρωθεί, αλλά ήδη υπάρχουν σχέδια ώστε να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε τους Αφγανούς αστυνομικούς σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση το ανεξάρτητο δικητήριο τοπικών, τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούμε να το ελέγξουμε γιατί είναι πολύ δύσκολο να τοποθετούμε Ευρωπαίους εκπαιδευτές σε διάφορα κομμάτια και επαρχές της χώρας. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά λεπτομερή προγράμματα που ήδη έχουν ξεκινήσει σε διάφορους τομείς, είτε είναι η εθνική κυβέρνηση, είτε είναι είτε είναι η στατικική κατά των ναρκωτικών κτλ. Είναι Πολύ δύσκολο λοιπόν να δούμε ποια είναι ακριβώς η ευρωπαϊκή στρατηγική δεδομένου των ποσών για τα οποία μιλάμε σε σύγκριση με άλλες χώρες και θεσμούς και δεδομένου της τεράστιας δομής προγραμμάτων δωρητών που έχουν ήδη συμφωνηθεί με τους ίδιους τους Αφγανούς. Και τα κεντρικά προγράμματα, αν βγάλουμε την ISAF, είναι η Αφγανική Στρατηγική Ανάπτυξης, η στρατηγική η ειρηνευτική, η στρατηγική για την δικαιοσύνη. Αυτά όλα υπάρχουν ήδη. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα πλογίσουμε ανάμεσα στις ίδιες υπάρχουσες στρατηγικές. Ευχαριστώ. Τώρα για να συνοψίσει ο κύριος Αρλάκη. Δύο παρατηρήσεις να κάνω για τα όσα είπε ο κύριος Κασουλίδης και οι υπόλοιποι. Το θέμα της προσέγγισης στρατηγικής είναι στην ουσία τυπικό, είναι μόνο ονομαστικό. Λέει η έκθεση νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν. Υπάρχουν ένα-δυο τροπολογίες που λέει ότι δεν είναι προσέγγιση αλλά στρατηγική. Ούτως ή άλλως σημασία δεν έχει το όνομα, το πώς θα το ονομάσουμε. Νομίζω πως ο τίτλος δεν μπορεί να αλλάχτεί. Ρώτησα από την, ε, τις της Επιτροπής μας και είπαν ότι... Ε, είναι λίγο περίπλοκο, πάση περιπτώσει. Έτσι κι αλλιώ δεν έχει νόημα, δεν έχει σημασία. Ούτε πρέπει να χρονοτριβούμε, να καθυστερούμε συζητώντα το όνομα. Συμφωνώ ότι η έκθεση ακολουθεί την φιλοσοφία, τη ε, εγώ πήγα στο Αφγανιστάν, το συζήτησα με τους Αφγανούς και πραγματικά με εντυπωσίασε το ότι συμφώνησαν με το 90% των όσων τους έλεγα. διότι η στρατηγική αυτή είναι πολύ, πολύ έξυπνη. Δηλαδή, μέσω της ε, στρατηγικής κατασκοπίας να καταλάβουμε το, και να αναλάβουμε το θέμα της, της αντίστασης, της αντιπολίτευσης. Προσπάθησαν να το δεχτούν όλα. Το βασικό ζήτημα είναι ο πληθυσμός. Μου είπαν, αρχίσαμε προσπαθώντας να καταλάβουμε γιατί χάσαμε την υποστήριξη του πληθυσμού και συμπεράναμε πως οι επικρίσεις ε, για μας, τον τρόπο με τον οποίο εμείς ε, διεξάγουμε τις επιχειρήσεις ε, επιτόπου, απομάκρυνε τον πληθυσμό λόγω των θυμάτων των αμάχων. Συμφωνούμε. Και ο Κρίσταλ προσωπικά είπε ότι στόχος μας είναι να έχουμε μηδενικές, μηδεν, θύματα άμαχους. Τον άκουσα με τα αυτιά μου τα ίδια να λέει στον, στους δικούς του ότι αυτή θα πρέπει να είναι η φιλοσοφία του τρόπου με τον οποίο παρεμβαίνουν επιτόπου. Εκτιμώ λοιπόν που βάζετε αυτήν την στρατηγική εικόνα εδώ στην έκθεση και δέχομαι την τροπολογία σας για αυτό το θέμα. Μία σύντομη παρατήρηση για τη δήλωση της Επιτροπής. Η έκθεση δεν θέλει ούτε ένα ευρώ παραπάνω για την στρατηγική αυτή. Κατά τη γνώμη μου αυτό που κάνει η Ένωση και τα κράτη-μέλη ήδη είναι αρκεί και περισσεύει. Δεν χρειάζονται παραπάνω χρήματα. Όχι, πρέπει απλώς να εξορθολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο δαπανούμε τα χρήματα. Το γεγονός ότι 80% αυτών των χρημάτων δεν φτάνει καν στον αφγανικό λαό, θα πρέπει να αρχίσετε να το εξετάζετε σοβαρά. Έχουμε στην Ένωση 200% της ενίσχυσης πάει στους διάφορους συμβούλους. Μα είναι υπερβολικό αυτό. 5-6% επισήμως αφορά την ασφάλεια. Έχουμε κόστος λειτουργίας υπερβολικό. Φτάνουμε δηλαδή στο 30% μίνιμουμ που δεν φτάνει καν μέχρι το Αφγανιστάν. Συγκρίνεται τι έκανε η Βραζιλία τα τελευταία 8 χρόνια, τι έκανε ο Λούλα <coughs> με τα ίδια χρήματα που δώσαμε όλοι εμείς στο Αφγανιστάν. 24 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βραζιλία βγήκαν από τη φτώχεια με αυτά τα χρήματα. Είχαν αυτά τα χρήματα τεράστιο αντίκτυπο στο Αφγανιστάν μετά από 8 χρόνια με τη δαπάνη των ίδιων χρημάτων έχουμε περισσότερους στόχους. Εξορθολογισμός λοιπόν των δαπανών και εξάλληψη του βάρους ε, της γραφειοκρατίας και όλα αυτά. Υπάρχουν και συμβολές των συναδέλφων που ζητούν καλύτερη ενημέρωση προς εμάς για το τι ακριβώς γίνονται τα χρήματα αυτά. Τεράστια προσπάθεια γίνεται για τη συλλογή των στοιχείων, γιατί είναι ένα πολύ συνεκτικό σύστημα. Ναι, ε, θα πρέπει μάλλον να γίνει ένα συνεκτικό σύστημα. Μα μάθουμε από του Αμερικανού. Αυτοί έχουν ένα σύστημα με αναφορέ. Μπαίνει κανεί στο ίντερνετ και σε δύο ώρε ξέρει τι δαπανάουν, πού, πώ και γιατί. Και όλα τα σχετικά έγγραφα του Κογκρέσου είναι διαθέσιμα. Ε, μπορεί κανείς να έχει όλα τα στοιχεία. Εγώ προσπαθώ μήνες για να βρω κάποια βασικά στοιχεία για να δω τι ακριβώς κάνουμε εμείς στο Αφγανιστάν από την Ένωση. Από τα κράτη-μέλη δεν υπάρχει περίπτωση να μάθει κανείς τι δαπανούν και σε τι. Προσπάθησα με τη χώρα μου. Αδύνατον. Γιατί το πώς δαπανούνται τα ιταλικά χρήματα εκεί είναι θαμμένο σε διάφορες γραμμές του προπολογισμού. Είναι σχεδόν αδύνατον να ξέρει κανείς τι γίνονται 700 εκατομμύρια ευρώ που κοστίζει η Ιταλική αποστολή στο Αφγανιστάν. Αδιακρίτως σε στρατιωτικά και πολιτικό σκέλος. Σε πάση περιπτώσει πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Εμείς στο Κοινοβούλιο και οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον να ξέρουν πώς δαπανώνται τα λεφτά τους με ξεκάθαρο και κατανοητό τρόπο. μόνο το τμήμα της έκθεσης που λέει κάποιες λεπτομέρειες για αυτή τη στρατηγική είναι τα ναρκωτικά. Γιατί έχουμε κάποια στοιχεία. Μετά από δέκα χρόνια δεν υπάρχει εθνικό πλάνο εξάλληψης των ναρκωτικών από το Αφγανιστάν. Το Υπουργείο κατά των Ναρκωτικών. Επισκέφθηκα το Υπουργείο, μίλησα με τους αρμοδίους κτλ. Αλλά δεν είναι σε θέση να δώσουν οτιδήποτε που να έχει σημασία η ε, νεπάρκεια και η διαφθορά βασιλεύουν, άρα δεν ε, έχει νόημα να συζητά κανείς με αυτούς. Πρότεινα να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο με, με, σώμα στο οποίο να συμμετέχουν αυγανοί. με επικεφαλής κάποιον όμως που να είναι αξιόπιστος με ένα σαφές πρόγραμμα πέντε χρόνων για να δούμε ποιε θα μπορούσαν να είναι εναλλακτικέ καλλιέργειες, χρησιμοποιώντα νέε νέες σπορές και νέε ευκαιρίε που υπάρχουν εδώ και μερικά χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα μέχρι ότου να φτάσει ω εδώ ο Υπουργό. Σας ευχαριστώ όλους όσους ήσασταν εδώ και συμμετείχατε σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Well, welcome to this uh, joint meeting. Uh, Καλώς ορίσατε. Σας καλωσορίζουμε από κοινού με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Έχουμε την τιμή να υποδεχόμαστε σήμερα εδώ την ε, εξοχότητά του, τον κύριο Μαχμούτ Σαντ Μεχμούτ Κερεσί, Υπουργό Εξωτερικών του του ε, Πακιστάν συνοδεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών και Οικονομίας, ε, ο γερουσιαστής Ιέντα Ουκραϊμάμ και ο πρέσβη Τζαλίλ Λαμπά Αντιλανή που είναι επίσης παρόν εδώ. Ε, να σας θυμίσω ότι έχουμε κάποιες σε ψηλού επίπεδο επισκέψεις ε, κατά τη διάρκεια αυτής της ε, θετίας, πολύ καλές ευκαιρίες για την ανταλλαγή απόψεων για μια περιοχή που είναι μεγάλο ενδιαφέροντος για τη Δυτική Ευρώπη, την Ένωση και όχι μόνο. Θα έλεγα ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακιστάν είναι εξαιρετική σημασία. Θα ήθελα να εκφράσω εξ ονόματο όλων ε, των παρόντων εδώ που αντιπροσωπεύουμε τις πολιτικές μας ομάδε, τη μεγάλη μας ε, συμπάθεια προς το λαό του Πακιστάν μετά από τις ε, πλημμύρες, τις καταστροφικές που δοκίμασαν την ε, χώρα σας. Ε, ξέρω πως αύριο θα συζητηθεί η συζήτηση και το θέμα θα είναι και πάλι στην ημερήσια διάταξη όταν θα συζητήσετε με την ΥΠΑ το εκπρόσωπο Άστον και την πρόεδρο της Επιτροπής και θα ήθελα να σας πω και ξέρω πως στην παρουσίασή σας θα τα θίξετε αυτά τα σημεία, αλλά θα ήθελα να σας εξοικειώσω με τα δικά μας ε, ενδιαφέροντα που σχετίζονται με τα πολιτικά ζητήματα όπως είναι οι σχέσεις με την Ινδία, και ιδιαιτέρως την κατάσταση στο Κασμίρ, η περιφερειακή σταθερότητα γενικότερα, ιδιαίτερα το ρόλο του Πακιστάν στην αναζήτηση της συμφιλίωσης του Πακιστάν, αγώνας κατά το εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας και φυσικά ανθρώπινα δικαιώματα. Με όλα αυτά λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εξοχότητά σας, ε, ώστε στη συνέχεια οι συνάδελφοι της Επιτροπής μας και της Αντιπροσωπείας μας να έχουν την ευκαιρία να πάρουν το λόγο και να μπορέσουμε να έχουμε και ένα κομμάτι χρόνου για ερωταπαντήσεις. Ε, ε μας είπατε ότι, έχετε κάποιο χρόνο στη διαθεσή σας και αυτό φυσικά θα το λάβουμε υπόψη ε, και μέσα στο πλαίσιο του κανονικού μας ωραρίου εργασίας. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντίβα, Πρόεδρε της ε, Επιτροπής ε, Ανάπτυξης, κυρία Λάμπερτ, Πρόεδρε της ε, Αντιπροσωπείας για την Ανατολική Ασία. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα σα που μου δώσατε την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας κάποιες απόψεις για τα θέματα που ε, ήδη αναφέρατε. Ο πρόεδρος μου είπε ότι η τελευταία επίσκεψη Πακιστανού εδώ ήταν ο πρώην πρόεδρός μας και ότι πολύ καυτά ερωτήματα του θέσατε και δύσκολα. Οπότε, επειδή είπα ότι έχω χρόνο στη διάθεσή μου, σας δίνω και μεγάλη, ε, την ευκαιρία να με δυσκολέψετε και εμένα. Να σας πω, λοιπόν, δύο λόγια για τις απόψεις του Πακιστάν και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πολύ σημαντικές. Είχαμε την επιθυμία να αναβαθμίσουμε τη σχέση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ένωσης και Έχουμε επίσης μεγάλη διασπορά στην Ευρώπη. Πολλά συμφέροντα λοιπόν έχουμε εδώ στην Ευρώπη. Και βεβαίως από δική σας πλευρά, από ευρωπαϊκής πλευράς υπήρξε ζωηρή ανταπόκριση στη δική μας επιθυμία. έχετε δείξει εκτίμηση για την προσπάθεια που καταβάλει το Πακιστάν στην καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της ε, τρομοκρατίας και αντικατοπτισμός. Αυτό ήταν οι διασκέψεις κορυφής που είχαμε την περασμένη χρονιά και φέτος και είμαστε, είναι ένα ποιοτικό άλμα στη σχέση μας το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερος. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω ως μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Επιτροπής Ανάπτυξης για την έκφραση αλληλεγγύης που δείξατε με το λαό του Πακιστάν, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των άνευ προηγουμένων πλημμυρών που αντιμετωπίσαμε. Όπως όλοι γνωρίζετε, καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν τη χώρα μας, επηρεάζοντας την ζωή 20 εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι αναγκάστηκαν να μετατοπιστούν εσωτερικά, να διασωθούν, να βοηθηθούν με κάποιο τρόπο. Ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα ήταν απαραίτητη και την προσέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπλέον η συνένεση που δημιουργήθηκε στην άτυπη συνεδρίαση με τους Υπουργούς Εξωτερικών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνέχεια, ώστε να δοθεί πλήρη ε, στήριξη στην οικονομική σταθερότητα του Πακιστάν. Αυτά είναι βήματα που εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα στο Πακιστάν και που έστειλαν ένα ε, πολύ θετικό μήνυμα στο λαό του Πακιστάν που είναι εταίροι σας ε, στην αγώνα τα του εξερμισμού και της τρομοκρατίας. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν παρουσία στην ε, περιοχή και φυσικά ενδιαφέρεστε και για την ασφάλεια των Ευρωπαίων που βρίσκονται στην περιοχή. Ήθελα να σας μιλήσω για την συνένεση στην οποία φτάσαμε ε, ο δημοκρατικά εκλεγμένος συνασπισμός, ε, κυβερνητικός συνασπισμός του Πακιστάν. Το Πακιστάν ήταν ε, σύμμαχος του ΝΑΤΟ της Ευρώπης και τον ΙΠΑ στον, ε, στο Αφγανιστάν σε αυτόν τον αγώνα κατά του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας. τα στρατεύματά μας είχαν ε, συμμετέχει. Αυτό που μας έλειπε όμως ήταν η πολιτική ιδιοποίηση αυτού του αγώνα. Και αυτό που έκανε η εκλεγμένη κυβέρνηση είναι ότι έδωσε αυτή την πολιτική ιδιοποίηση αυτού του αγώνα. Για να γίνει αυτό ε, χρειάστηκε να γίνει μια συζήτηση εντό και εκτός κοινοβουλίου και τελικά καταλήξαμε πως όλοι έπρεπε να συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγώνα σαν να ήταν ο δικός μας και αυτό καταφέραμε και το αποτέλεσμα ήταν πως οι ενέργειές μας τα τελευταία δυόμιση χρόνια ήταν πιο ε, ουσιαστικές και πιο επιτυχείς ως, εκ τούτου και ο κόσμος αυτό το αναγνωρίζει. Τώρα βέβαια υπάρχει το τίμημα, το οικονομικό το οποίο πληρώσαμε, αναπόφευκτο είναι αυτό. Κανένας δεν μπορούσε να το προβλέψει αυτό. Ε, ε, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της ευθυγράμμισης είναι προφανής. Εκροή κεφαλαίων, έλλειψη επενδύσεων και λόγω της ισχύωσης κατάστασης ο, δεν είναι ο κόσμος πρόθυμος να ταξιδέψει εκτός της χώρας να συναντήσει τους πελάτες του. Αυτό είναι τίμημα το οποίο χρειάστηκε να καταβάλουμε. Και φυσικά κληρονομήσαμε μια αρκετά δύσκολη οικονομική κατάσταση, διότι όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση, όλοι οι μακροοικονομικοί μας δείκτες δεν ήταν τόσο σταθεροί όσο θα έπρεπε. Επιπλέον μας χτύπησε η παγκόσμια ύφεση όπως σε όλους. Αύξηση των τιμών του πετρελαίου και ούτω καθεξής. Οι οικονομικές μας δυσκολίες λοιπόν πολλαπλασιάστηκαν καθώς άρχισε τη θητεία της νέα δημοκρατική κυβέρνηση. Εμείς τώρα προβήκαμε σε διάφορα δύσκολα, οδυνηρά πολιτικά βήματα, αυξάνοντας τους δασμούς, αναστέλλοντας ε, ενισχύσεις, το αποτέλεσμα ωστόσο ήταν ότι μπορέσαμε σε μεγάλο βαθμό να σώσουμε τους επιδεινούμενους οικονομικούς δείκτες, μπορέσαμε να μειώσουμε ε, τον πληθωρισμό, το κρατικό μας έλλειμμα, το ποσοστό των ανθρώπων που ζούσαν κάτω από το επίπεδο της στόχης, δεν αυξήθηκε, ωστόσο οι πλημμύρες δεν βοήθησαν. Τώρα πρέπει να διπλασιάσουμε την προσπάθεια για να επανέλθουμε σε την προηγούμενη μας κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, το Πακιστάν ανακουφίστηκε πριν από ένα χρόνο από τη πλευρά της Ευρώπης λόγω αυτού του σχεδίου GSP+, δηλαδή του καθεστώτος προτιμούμενου ε, προτιμησιακού μάλλον καθεστώτος, ε, πράγμα που έδωσε μεγαλύτερη πρόσβαση και ε, Ωστόσο είδαμε μια πτώση των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν αυτές μειώνονται αυτό μας ε, ζημιώνει σε μεγάλο βαθμό γιατί είστε ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς μας εταίρους. Εάν θέλετε να μας βοηθήσετε να καταπολεμήσουμε όμως τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία, ένα τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο είναι να γίνει σταθερό οικονομικά το Πακιστάν. Ε, όταν είμαστε εμεί σταθεροί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της στόχης και όταν είμαστε οικονομικά σταθεροί θα μπορείτε να επενδύσετε σε τομείς που έχουν παραμεληθεί στο παρελθόν όπως υγεία, παιδεία, αν όμως έχουμε να κάνουμε με τον εξτρεμισμό μακροπρόθεσμα, η μακροπρόθεσμη λύση στον εξτρεμισμό είναι η παιδεία. Πρέπει ο κόσμος να εκπαιδευτεί, να καλλιεργηθεί, γιατί έχουμε δει ότι οι τομείς, οι περιοχές όπου ο αναλφαβητισμός και η φτώχεια βασιλεύουν, εκεί είναι η πηγή για τους εξτρεμιστές. Εκεί είναι το κατάλληλο έδαφος, γόνιμο έδαφος για να μπορέσουν να στρατολογήσουν οι εξτρεμιστές. Η πρόσβαση λοιπόν στην αγορά θα είναι πολύ χρήσιμη, θα βοηθήσει την οικονομία και είμαι ευτυχής που εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο. Η Υπουργοί σε άτυπη συνάντηση συμφώνησαν ότι αυτό θα είναι χρήσιμο για το Πακιστάν, ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο και ότι θα ε, στηρίξει και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πακιστάν. Να σας μιλήσω μισό λεπτό για την εσωτερική κατάσταση, για τις εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα. Από τότε που η κυβέρνησή μας ανέλαβε καθήκοντα, υπήρξαν διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες. Καταρχήν, εκλογές αναγνωρίστηκε ότι διεθνώς και σε εθνικό επίπεδο ήταν αξιόπιστες και δίκαιες και τα αποτελέσματά τους έγιναν αποδεκτά. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση με την οποία συνομιλείται σήμερα είναι μια δημοκρατικά εκλεγμένη νόμιμη κυβέρνηση σε αντίθεση με την κυβέρνηση την οποία είχατε ε, ως συνομιλητή παλιότερα. Εμείς, έχοντας υπόψη τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ε, ακολουθούμε μια πολιτική συμφιλίωσης. Και γι' αυτό στο, οι πολλοί από τους ε, αντιπάλους των παρελθόντων συνεργάζονται ως ε, εταίροι τους στο κυβερνητικό συνασπισμό σήμερα. Γιατί οι προκλήσεις μας είναι τεράστιες και πρέπει να μπορέσουμε να αντλήσουμε από τους πόρους που έχουμε στη θέση μας για να τις αντιμετωπίσουμε. Έχουμε λοιπόν κυβερνητικό συνασπισμό στο κέντρο, αλλά και στις τέσσερις ε, ε, ομοσπονδιακές περιφέρειες της χώρας. Όταν λαμβάνουμε καθήκοντα, οι νομικοί διαδήλωναν για την αποκατάσταση πολλών από τους δικαστές που είχαν απολυθεί από το προηγούμενο καθεστώς και καταφέραμε να αποκαταστήσουμε την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Σήμερα μπορούμε να πούμε πως στο Πακιστάν έχουμε ένα ανεξάρτητο και αξιόπιστο δικαστικό σώμα. Έπειτα θα έλεγα πως είναι η πρώτη πολιτική κυβέρνηση που δείχνει μεγάλη υπομονή και επιτρέπει την ανεξαρτησία των ΜΜΕ ηλεκτρονικών και άλλων. Διότι αναγνωρίζουμε ως δημοκράτες πως αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία. Αν κανείς πιστεύει στη δημοκρατική κουλτούρα και στις δημοκρατικές αρχές, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν ανεξάρτητα Ε. Και αυτό πάλι βοηθά ώστε πολλές περιοθωριοποιημένες, περιοθωριοποιημένα κομμάτια της κοινωνίας να έχουν πια μια φωνή, να παίζουν το επίσης ρόλο ελεγκτή, ε, παρέχουν διαφάνεια στο σύστημα, πολύ θετικές εξελίξεις και αυτές. Έγιναν επίσης συνταγματικές αλλαγές. Αλλαγές στο Σύνταγμα Ιδιαίτερα στο 17ο άρθρο που μεταφέρει την ισορροπία από την κοινοβουλευτική δημοκρατία που είχαμε με ένα υβρίδιο, δεν ήταν ούτε, ούτε κοινοβουλευτική δημοκρατία ούτε προεδρικό σύστημα. Σήμερα, μέσω μια ανοιχτή συζήτηση, καταφέραμε να θέλουμε δύο τρίτα πλειοψηφία για οποιαδήποτε αλλαγή στο Σύνταγμα. Εμεί ω πολιτικό κόμμα δεν το είχαμε αυτό το ποσοστό. Άρα λοιπόν έγινε μια πολύ ζωηρή συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Και το, η, συντα, η συνταγματική μεταρρύθμιση που προτάθηκε από την κυβέρνηση εγκρίθηκε ομόφωνα. Όχι μόνο από τα δύο τρίτα της πλειοψηφίας, Και έτσι μπορέσαμε να αφαιρέσουμε όλες τις τρευλώσεις που υπήρχαν στο Σύνταγμα παλαιότερα. Μια άλλη σημαντική πολιτική εξέλιξη στο Πακιστάν ήταν ότι Υπήρξε μια μετακίνηση λοιπόν από το κέντρο, από την κρατική κυβέρνηση προς τις επαρχίες, προς τις περιφέρειες. Προσπαθούμε να βρούμε, μάλλον λειτουργούσαμε με μια ad hoc ρύθμιση τα τελευταία 19 χρόνια. Εμείς φτιάξαμε μια Εθνική Κυβέρνηση ε, Επιτροπή Οικονομίας και έχουμε διαπραγματευτεί με τις επαρχίες και την κεντρική κυβέρνηση ένα νέο ε, ε, εθνικό οικονομικό σύστημα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιο, πιο συντονισμένα. Υπάρχουν, υπάρχει σαφής ε, διαχωρισμός για το ποια έσοδα πάνε στην κρατική, κεντρική κρατική κυβέρνηση και ποια έσοδα πάνε στις επαρχίες και στις περιφέρειες. Πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή. Επίσης δημιουργήσαμε ένα νέο φόρουμ. Ένα φόρουμ ε, ε, για συζήτηση. Εκτός από τις υπουργικέ δηλαδή διασκέψεις. Αυτό δημιουργήθηκε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε φιλίες με όλη την Ευρώπη και με ολόκληρο τον κόσμο, με δημοκρατικές χώρες, δημοκρατικές αρχές να έχουμε ένα φόρουμ το οποίο να μπορεί να κατανοήσει τα θέματά μας και να κατανοήσουμε και εμείς ποιες είναι οι ανησυχίες των εταίρων μας. Σαν φίλοι να τα αντιμετωπίσουμε και νομίζω πως αυτό το φόρουμ γίνεται σιγά σιγά πολύ ενδιαφέρον. Πολλές πολιτικές εξελίσσονται. Για παράδειγμα, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ενεργειακού ελλείμματος και μέσω αυτού του φόρουμ αναπτύξαμε μια νέα έκθεση για την ενέργεια που εγκρίθηκε από αυτό το φόρουμ και συζητώνται και άλλα θέματα. Δεν χρειάζεται να σας τα πω όλα, όλες τις λεπτομέρειες, αλλά έτσι δημιουργήσαμε έναν διπλωματικό χώρο για τη χώρα μας που νομίζω είναι πολύ χρήσιμος. Τώρα, για τα θέματα των σχέσεών μας με την Ινδία που με ρωτήσατε κι εσείς Πρόεδρε. Για ε, το Πακιστάν με την Ινδία, ξέρετε, έχουμε κρεμότητες μεταξύ μας από το 1947, από τότε που ε, δημιουργηθήκαμε ως χώρες, υπάρχουν συγκρούσεις, έχουμε υπάρξει και πόλεμοι, ένοπλες σειράξεις αρκετέ φορές, αλλά αυτή η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση είναι της άποψης ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε ως καλοί γείτονες. Και οι δύο πλευρές είναι υπέρ της ρύθμισης των θεμάτων. Υπάρχουν θέματα, δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε ή να τα αποκρύψουμε, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε για έναν μηχανισμό επίλυσης και ο καλύτερος μηχανισμός επίλυσης είναι μια ειρηνική λύση μέσω διαπραγμάτευσης. Μόνο διάλογος μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε και αυτό το έχουν συμφωνήσει δύο πρωθυπουργοί και δύο υπουργοί εξωτερικών έχουν αναλάβει το έργο του να προχωρήσουν και να γεφυρώσουν το χάσμα εμπιστοσύνης, να δημιουργήσουν δηλαδή εμπιστοσύνη και να προχωρήσουμε σε όλα τα εκκρεμή θέματα γίνονται διαπραγματεύσεις, ε, ε, μάλλον αναστάλθηκαν για λίγο καιρό. Ευτυχώς και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν. Ο Υπουργός μας ήταν στο Πακιστάν τον Ιούλιο. Είχαμε μια πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων. Προσεκλήθην στην Ινδία να επισκεφθώ το Δελχή Έχουμε ένα πακέτο προσυζήτηση που μπορεί να είναι χρήσιμο και για τις δύο πλευρές. Προοδευτικό. Εγώ προσωπικά πιστεύω πως όλα ένα και περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι ο κόσμος θέλει τη ρύθμιση, τη σταθεροποίηση, την ειρήνη στην περιοχή. Το Κασμίρ είναι θέμα. Ε, ναι, καθένα ήταν πρόβλημα. Τον τελευταίο καιρό αναφέρεται διαρκώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης λόγω των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί, αλλά ποιο είναι το θετικό στοιχείο ότι το Πακιστάν μπορεί να το ισχυριστεί αυτό, αλλά όχι μόνο το Πακιστάν. Η διεθνής κοινή γνώμη και η κοινή γνώμη στην Ινδία, οι διανοούμενοι, οι ακαδημαϊκοί, το Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά να γνωρίζουν ότι αυτή η ανησυχία, αυτή η αταξία είναι ε, γενής εκεί στη φύση της και ότι δεν ε, τα ρίχνουν όλα στο Πακιστάν. Ναι, καθένα εμεί αυτό κάναμε. Εμεί τα ρίχναμε στου Ινδού, οι Ινδοί σε εμά και πάει λέγοντα. Αυτή τη στιγμή και, τα, και οι δύο πλευρέ αναγνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα και θέλουν να βοηθηθούν, να, να βοηθήσουν αλλήλους να αντιμετωπίσουν αυτές τις πραγματικότητες. Αυτή είναι η πρόκληση λοιπόν. και θέλουμε η ηγεσία του Κασμίρ να μπει μέσα στην ομάδα των διαπραγματεύσεων, το συζητήσουν ώστε τα ζητήματα να λυθούν θετικά, με πολιτικό τρόπο. Το πρόβλημα είναι πολιτικής φύσης. Και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργό Μαν Μονσίνκ το αναγνώρισε αυτό. Είναι πολιτικό το ζήτημα και χρειάζεται πολιτική λύση. Και αν υπήρξε εδώ μια κίνηση, το Πακιστάν Φυσικά και θα ήθελε η κατάσταση στο Κασμίρ να βελτιωθεί. Για το Αφγανιστάν. Το τελευταία δύο χρόνια και μάλλον το και του τελευταίου έτους έχει αναγνωριστεί ότι οι σχέσεις με το Αφγανιστάν έχουν βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν δαχτυλοδείχνουμε πια ένα στον άλλον, δεν αλληλοκατηγορούμεθα. Συνομιλούμε. Περισσότερο από παλιότερα σε όλα τα επίπεδα, σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο στατιστικό σε επίπεδο ε, υπηρεσιών. Υπάρχουν περισσότερες κοινοβουλευτικέ αντιπροσωπείες. Μόλις υπογράψαμε μια νέα ε, μεταβατική συμφωνία με διέλευση με το Πακιστάν, δύο συμφωνίες για διμερή συνεργασία με το Πακιστάν που ξεπερνούν τις προηγούμενες μας ε, συμφωνίες, θέτουν τα θεμέλια για μια ε, συνεργασία με το Αφγανιστάν έχουμε στηρίξει όλες τις διεθνείς προσπάθειες για σταθερότητα και ειρήνη στο Αφγανιστάν. Και τελευταία απόδειξη ήταν η διάσκεψη του Λονδίνου, όπου Όλοι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών ήταν παρόντες και το Πακιστάν ενέκρινε και στήριξε την στρατηγική της κυβέρνηση Ομπάμα. Επίσης, αναλαμβάνουμε κάποια προγράμματα που πιστεύουμε ότι θα βελτιώσουν τη συνεργασία με το Αφγανιστάν να αναδομήσουμε, να, μάλλον, να αναβαθμίσουμε τους, ε, το δικό και το σιδηροδρομικό μας δίκτυο προς το Αφγανιστάν και επίσης προσφέραμε να βοηθήσουμε στην διαδικασία συμφιλίωσης. Προφανώς θα πρέπει να είναι αφγανική βασικά η προσπάθεια και θα πρέπει αυτήν να την ιδιοποιηθεί και να την, της ηγηθεί το ίδιο το Αφγανιστάν. Αλλά εμεί μπορούμε να βοηθήσουμε. Γιατί η διαφορά του Πακιστάν είναι ότι σήμερα υπάρχει αναγνώριση ότι δεν μπορεί να υπάρχει σταθερότητα και ειρήνη στο Πακιστάν αν δεν υπάρχει ειρήνη και, και σταθερότητα και στο Αφγανιστάν. Δηλαδή τα συμφέροντά μας είναι αλληλένδετα. Και αυτό έχει επιφέρει αλλαγή στον τρόπο σκέψης και έχει ε, φέρει πιο κοντά τις δύο χώρες. Δουλεύουμε καλύτερα και κατανοούμε αλλήλως καλύτερα. Μιλήσατε για τον αγώνα κατά του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας και εδώ ήμασταν επιτυχείς στην μετατροπή της κοινή γνώμης του Αφγανιστάν κατά του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας. Σήμερα η κοινωνία των πολιτών σήμερα εκτός από ορισμένα ακραία θρησκευτικά κόμματα. Ε, η, βασικά όμως η ευρεία πολιτική συνένεση είναι κατά του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας. Και έχει σημειωθεί πρόοδος. Εμείς τώρα είμαστε μια πολιτική κυβέρνηση, είμαστε υπόλογοι στο λαό. Πρέπει να πάμε κάποια στιγμή στις κάλπες πάλι. Και σήμερα έχουμε ανεξάρτητα με μη ε, ελεύθερα, με πολύ... έχουμε ανεξάρτητο δικαστικό σώμα όπως είπα και... Κυβερνά μια γυναίκα. Η Μπενιζέ Πότο. Αυτή, που κυβερνούσε ήταν αυτή, όπως το ξέρετε, που ήταν πολύ δημοκράτης, θέλουν να δώσουν ε, το κόμμα ε, τα δικαιώματά τους στις μειονότητες, να τις αναγνωρίσουν, να τους δώσουν τη σωστή τους θέση, να αντιμετωπίσουν τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σήμερα συμφωνήσαμε και εμείς πια στις 37 συμβάσεις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι όπως ξέρω πολύ σημαντικές και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, γι αυτό το... και σε αυτό το επίπεδο λοιπόν υπήρξε πρόοδος. Εν κατακλείδη λοιπόν θα έλεγα ότι ναι έχουμε προκλήσεις, έχουμε δυσκολίες. Δεν λέω ότι όλα τα έχουμε λύσει. Όχι, πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν. Αλλά έχουμε αρχίσει πια να προχωρούμε μπροστά σε όλους τους τομείς που είναι ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Πακιστάν. Σήμερα λοιπόν έχουμε θεσπίσει τα θεμέλια Έχουμε θέσει τα θεμέλια για μια μακρά ε, εταιρική σχέση, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πολύ σημαντική για το, για το Πακιστάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακαλέσω τώρα την κυρία Λάμπερτ να λάβει το λόγο και τον κύριο Ντέβα και μετά ε, όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι που έχω το όνομα τους εδώ στον κατάλογο. Παρακαλώ κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Υπουργέ για την εκτενέστατη αυτή παρουσίαση και εξήγηση των όσων συμβαίνουν στο Πακιστάν μετά τις δημοκρατικές εκλογές ε, για τη Βουλή και το σχηματισμό της κυβέρνησης. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών, εκφράζουμε τα ειλικρινά μας συλληπιτήρια για τα όσα υπέστη ο λαός του Πακιστάν και τα συνεχιζόμενα προβλήματα που απορρέουν από τις πλημμύρες, ε, την εκτόπιση των πληθυσμών, αλλά και πριν τις πλημμύρες. Ίσως μία-δύο ερωτήσεις από πλευράς μου. Ε, το ένα ερώτημα έχει να κάνει με θέματα διεθνούς υποστήριξης για την ανοικοδόμηση μετά τις πλημμύρες. Και ένα θέμα που έχει ανακύψει είναι η λογοδοσία και η διαφάνεια της διαχείρισης των γοδηλίων που ρέουν τώρα προς τη χώρα. Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς ε, το διαχειρίζεστε αυτό. Και επίσης από την κοινοβουλευτική σκοπιά Ανησυχεί ο κόσμος στο Πακιστάν, από ό,τι φαίνεται, για το εξή. Τα δημοκρατικά εκλεγμένα σώματα είναι αόρατα για τους πολίτες ή δεν, φάνηκαν, δεν έκαναν αισθητή την παρουσία τους ε, τη στιγμή των πλημμυρών. Εσείς πώς θεωρείτε ότι επηρεάζει την αίσθηση του κοινού και της κοινή γνώμης για το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση. Και ακόμα ένα ερώτημα και σε σχέση με αυτό αλλά και γενικότερα με την ανάπτυξη. Ποια πρόοδος έχει γίνει ως προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ προφανώς για το τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο, τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Αλλά αυτό πώς διαχέεται ε, επιτόπου γιατί η οικονομική ανάπτυξη θα έρθει από την οικοδόμηση και από το εκπαιδευτικό σύστημα κτλ. Τι προτείνετε λοιπόν για να ενισχυθεί η τοπική διακυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντίβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξοχότατε, Υπουργέ, κύριε Κιουρέση. Δεχθείτε παρακαλώ τα συλληπιτήρια της Επιτροπής Ανάπτυξης για την τραγωδία που έπληξε τη χώρα σας. 21 εκατομμύρια είναι εκτοπισμένοι και περίπου 11 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Ενώ εκατοντάδες, χιλιάδες είναι νεκροί. 400 εκατομμύρια ε, ευρώ έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ένωση και 150 εκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανθρωπιστική βοήθεια και μόνο. Η αναπτυξιακή βοήθεια είναι κάτι το οποίο ακόμα συζητείται. Ο Κάρλ Ντεχούχτ την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε 900 εκατομμύρια ευρώ ως διευκόλυνση για να μπορέσουν οι ε, εξαγωγές σας να ε, έρχονται στην Ένωση ε, ε, αδασμολόγητα με την, εξαίρεση, την περίεργη εξαίρεση των ε, προϊόντων, κυρίως λινά τραπεζομάντιλα, δεν ξέρω για ποιο περίεργο λόγο είναι αυτό. Όταν έπληξε το τσουνάμι της Σιλάνκα ήμουν εκεί στον 8ο όροφο και κοίταζα τι συνέβαινε ε, μπροστά στα μάτια μου και αυτό ήταν τρομερά τραυματική εμπειρία στη δική μου ζωή. Φαντάζομαι ε, ε, και εσείς τι εμπειρίες θα είχατε από τις πλημμύρες. Κάτι όμως ε, που λυπάμαι πάρα πολύ και δεν μπορώ να το απαντήσω και αντιμετώπισα πρόσφατα ήταν ε, το τσουνάμι χτύπησε την Ινδονησία ο απλός κόσμος μάζεψε στην Ευρώπη 4 δισεκατομμύρια δολάρια ε, ευρώ μάλλον ο απλός πολίτης ο καθημερινός πολίτης, όχι τα όργανα. Συνέλεξαν περίπου 5 δισεκατομμύρια ε, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Αν κάνουμε τώρα κάποιες συγκρίσεις, στο βαθμό που έχουν κάποια εγκυρότητα αυτές, 600.000 ήταν εκτοπισμένοι στη Σρι Λάνκα από το τσουνάμι και ε, πολύ λιγότεροι νεκροί ε, Στη δική σας χώρα ε, είπαμε 21 εκατομμύρια εκτοπίστηκαν και πολλοί έχασαν τις ζωές τους, πολύ περισσότεροι. Ωστόσο η παγκόσμια αντίδραση σε αυτό το φρικτό γεγονός ήταν ε, πιο περιορισμένη. Ο λαός της Ευρώπης δεν ε, συγκινήθηκε όπως στην περίπτωση της Ριλάνκα και της Ινδονησίας. Χρειάζονται δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων, μιλιούνια δολάρια και ε, ευρώ για να ξανασταθεί στα πόδια της η χώρα σας. Ωστόσο, δεν καταφέρατε να προκαλέσετε αυτή τη συμπόνια, τη συμπαράσταση ε, που γέννησε στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, ε, ας πούμε το τσουνάμι, άλλη φυσική καταστροφή, άλλη θεομηνία. Οι λαοί της Ευρώπης είναι καλοί άνθρωποι. Εγώ έχω περίπου 8 εκατομμύρια ε, ψηφοφόρους και συμμετέχω σε συνεδριάσεις και θυμάμαι ότι είχαν κάνει τρομερούς εράνους. Ε, έκλειναν ε, αίθουσες συνεδριάσεων, θέατρα, με καλούσα να μιλήσω και μάζευαν 500.000 στερλίνες μέσα σε ένα βράδυ. Εσείς πώς δεν έχετε φέρει στο πλευρό σας τους καθημερινούς πολίτες της Ευρώπης. Εντάξει τα θεσμικά όργανα, αλλά θα πρέπει και ο λαός να το κάνει δική του υπόθεση, να το αστερνιστεί. Ε, τι σας ε, ζητώ έτσι με αυτόν τον έμεσο τρόπο. Ξεκινήστε μια εκστρατεία για να συμπαρασύρετε και τους λαούς της Ευρώπης και να τους φέρετε στο πλευρό σας. Ε, για να συμμεριστούν και την ανθρωπιστική πλευρά και την προσπάθεια ανοικοδόμησης της χώρας. Ένα δεύτερο. Ίσως είναι ηρωνικό αυτό. Και πάλι κάνω τον παραλυσμό με τη Σιλάνκα, η οποία τα τελευταία χρόνια έζησε πραγματική κόλαση με τη τρομοκρατική οργάνωση εκεί. Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον ε, περασμένο αιώνα ξέρουμε ότι ε, Εκατό εκατομμύρια Ευρωπαίοι αλληλοσκοτώνονται και τώρα ε, συμμετέχουν μαζί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γάλλοι, Γερμανοί, Ιταλοί, Βρετανοί λαμβάνουν αποφάσεις κοινέ Το κοινοβούλιο αυτό ε, και ξεκινάει και αποφασίζει 80% της νομοθεσίας που αφορά το Σάσαξ και το Σάρι, την εκλογική μου περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει. Και ορισμένοι από εμά, το Συντηρητικό Κόμμα, δεν είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι με αυτή την εξέλιξη, είναι όμως γεγονός. και οι χρονολογίες είναι οι ίδιες. Ε, από τότε που επέκτησε την ανεξαρτησία της η Ινδία, το Πακιστάν και η Σρι Λάνκα έχουν περάσει τα ίδια χρόνια και στην Ευρώπη είδαμε τι έχει γίνει. Ενώ στην ε, υποήπειρο αυτή της Νότιας Ασίας ε, ακόμα μιλάμε για το 47 και για το 48 και στη Σρι Λάνκα το ίδιο. Μα πάνε τόσα χρόνια από τότε. Κοιτάξτε τι έκανε η Ευρώπη. Θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ο κόσμος προχώρησε. Και στην Νότια Ασία, στην παιδική μας περιφέρεια, δεν το έχουμε κατακτήσει αυτό. Έχουν δείξει το δρόμο οι Ευρωπαίοι. Έχουν ανοίξει το δρόμο για το πώς θα ζούμε όλοι εν ειρήνη. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Νομίζω γνωρίζετε ότι θα έχετε την ευκαιρία στη συνέχεια να απαντήσετε και μετά έχουν ζητήσει το λόγο πολλοί συνάδελφοι για να κάνουν ερωτήσεις. Αλλά πρώτα ο υπουργό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να αρχίσω από την κυρία Λάμπερτ. Ανθίξατε το θέμα της διαφάνειας στη χρήση ε, της οικονομικής βοήθειας που δίνεται στο Πακιστάν. Βεβαίως. Έχουμε αναγνώριση και επίγνωση του γεγονότος αυτού και κάνουμε βήματα ε, για να το αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την εξή σκέψη. Έγινε συζήτηση και ε, μάλιστα εκτεταμένη με τις ε, επαρχιακές κυβερνήσεις και τώρα έχει συσταθεί ένα συμβούλιο εποπτικό, εποπτικό συμβούλιο, 15 μελές μάλιστα, όπου συμμετέχουν συνταξιούχοι ε, ανώτατη δικαστική, συνταξιούχοι, ανώτατη ε, δημόσια υπάλληλη, κρατική λειτουργή και αξιοστέβαστα μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Είναι λοιπόν ένα σώμα το οποίο εποπτεύει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια για να ε, έχει την εμπιστοσύνη και ο κόσμος όλος αλλά και ο λαός του Πακιστάν ότι τα χρήματα πιάνουν τόπο. Οι και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε εγκαταστήσει μηχανισμούς, ελέγχους και ισορροπίες για να αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα ε, σωστά. Και παρακαλώ να μην έχετε κανένα φόβο ε, και καμία ανησυχία προκειμένου. Για το θέμα τώρα των δημοκρατικών θεσμών και των οργάνων που λέτε ότι δεν φαίνονται ή δεν έκαναν αισθητή την παρουσία τους όταν μας τύπησε αυτή η τρομερή θεομηνία. Μαθαίνετε βέβαια από τον τύπο ότι συμβαίνει, αλλά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όσοι επισκέφθηκαν τη χώρα ο διεθνή τύπο, δηλαδή, διεθνεί μη κυβερνητικέ οργανώσεις, διεθνείς ηθήνοντε, σήμερα δεν έχουν την ίδια αίσθηση εκείνη που επικρατούσε το παρελθόν, γιατί είδαν πραγματικά τι γίνεται επί τόπου και τις ε, τοπικές αυτοδιοίκησεις ε, συναντήθηκαν με μη κυβερνητικέ οργανώσει, δικέ μα με μέλη του Κοινοβουλίου που πηγαίνουν στο λαό. Εγώ βουλευτή είμαι κι εγώ και πρέπει να επανεκλεγώ. Θα πρέπει να απευθύνομαι στους ψηφοφόρους μου. Και αν δεν είμαι στο πλευρό τους, αν δεν τους συμπαραστέκομαι σε αυτή την αγωνία τους, ε, δεν βοηθάω και τον εαυτό μου. Δηλαδή, αυτή η εντύπωση που δημιουργήθηκε ε, ότι ε, απουσιάζουν οι δημοκρατικοί θεσμοί είναι στρεβλή. Βεβαίως στην αρχή όταν ε, ενέκυψε κάτι τέτοιο χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί με νέους θεσμούς. Χρειάστηκε να οικοδομηθούν ε, οι θεσμοί. Και αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αλλά όταν υπάρξει μια θεομηνία, ε, τρέχουν οι αρμόδιοι θεσμοί και οι αρμόδιοι φορεί να σώσουν τον κόσμο. Και έγινε αυτό σωστικά συνεργεία και με στρατιωτικού και με παραστρατιωτικού μηχανισμού και με πολιτικού μηχανισμού. Το, το ξέρουμε. Ε, αλλά τώρα έχει αναλάβει η εκάστοτε τοπική αρχή. Τώρα που μιλούμε για τη ανακούφιση για την παροχή ε, βοήθειας επίγουσας. Ποιος το κάνει αυτό, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι ε, ε, επαρχιακές διοικήσεις, αρμόδιοι για θέματα εκπαίδευσης, αλλά ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Παγκόσμια Τράπεζα, η Τράπεζα Ανάπτυξης, η Ασιατική, ε, που κάνουν κάποιες απογραφές ε, για να δουν τι βοήθεια χρειάζεται ο πληθυσμός. Όλα αυτά γίνονται σε τοπικό επίπεδο. Και να είστε βέβαιοι ότι τώρα έχουν αναλάβει και οι πολιτικοί ε, ενώ την πολιτική βοήθεια σε αντιπαράθεση και αντιδιαστολή με τη στρατιωτική. Και ένα άλλο στοιχείο που αναφέρατε ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό γιατί και εγώ ίδιος είμαι προϊόν ε, αυτής ε, της διοίκησης. Εγώ ήμουν ε, σύμβουλος ε, σε ένα τοπικό συμβούλιο, ε, δημοτικό συμβούλιο υπαρχιακό αν θέλετε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να Υπάρχει αυτή η διαδικασία και γίνεται για το Πακιστάν. Θα ήθελα να αναγνωρίσω όντω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε και σημαντικά βήματα προς την ορθή κατεύθυνση. Και θα πρέπει πάντα να αναγνωρίζουμε και τα θετικά που έχουν κάνει προηγούμενοι το προηγούμενο καθεστώ σε ό,τι αφορά την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και την εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων από το κράτος στις επαρχίες. αυτό έγινε από τις επαρχίες τώρα στην τοπική ε, αυτοδιοίκηση. Εμείς όμως ως κόμμα και ως κυβέρνηση θεωρήσαμε ότι πρέπει ακόμα περισσότερο να προχωρήσουμε και τώρα έχουμε με την 18η τροπολογία ε, στο Σύνταγμα δώσαμε περισσότερες εξουσίες από την κεντρική κυβέρνηση στη ε, περιφερειακή, την επαρχιακή προκειμένου και στη συνέχεια στην τελείω τοπική αυτοδίκηση. Και αυτό αφορά και θεσμικά ζητήματα αλλά και οικονομικά. Αυτό τον καιρό προσπαθούμε να ε, κάνουμε αυτή την τροποποίηση είναι θέμα που αφορά τις επαρχίες, οι οποίες νομοθετούν επίσης. Και τώρα θέλουν να ζητήσουν και εκλογές. Μάλλον είχαν την πρόθεση πριν τις πλημμύρες. Αλλά αυτό το θέμα των πλημμυρών νομίζω ανέβαλε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον στο προσεχές μέλλον δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές Και στο κάτω-κάτω από πού θα προέρθει η μελλοντική ηγεσία. Οι μελλοντικοί ηγέτες θα αναδυθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και η ιστορία της Νότιας Ασίας ευρύθη τέτοιων καταστάσεων. Έτσι έχουν αναπτυχθεί. Αρχής γενομένης ε, από την ίδρυση, ας πούμε, των κρατών. Ε, κύριε Ντίβα, αναφέρατε κι εσείς πολλά ζητήματα. Πρώτον, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Κατά τη διάρκεια των πλημμυρών ε, δεν είχαμε τόσα πολλά θύματα όπως στο σεισμό του 2005 που ήταν 80.000 οι νεκροί. Τώρα ήταν μόνο 1.700 οι νεκροί τα θύματα. Αλλά οι οικονομικές απώλειες είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με τους σεισμούς του 2005. Στη συνέχεια αναφερθήκατε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε γνώμονες που μας δίνουν τόσο μεγάλη οικονομική βοήθεια. Στη Γενέβη με τον ΠΟΕ θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, την προσπάθεια αυτή και ε, προσβλέπουμε στη δική σας υποστήριξη. Και τα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν λόγο και παρακαλώ να μας υποστηρίξετε. Ε, 900 εκατομμύρια ευρώ λέτε για ένα πακέτο. Ε, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Εμπορίου, ε, που μόλις συναντήσαμε, πρόκειται για 100 εκατομμύρια, όχι για 900 εκατομμύρια, όπως αναφέρετε εσείς. Το τρίτο που θέσατε είναι η παγκόσμια αντίδραση ε, στο, για τις πλημμύρε λέτε ότι ήταν κάπως μετριασμένη σε σχέση με την προηγούμενη. Κοιτάξτε, και εγώ ανησύχησα στην αρχή. Γιατί η διεθνή κοινότητα δεν ανταποκρίθηκε. Στη συνέχεια έμαθα από ανθρώπους που είχαν γνώση των πραγμάτων ότι είναι ε, διαφορετική η αντίδραση σε σεισμό και σε τσουνάμι από εκείνη των πλημμυρών. Γιατί τα θύματα δεν είναι τόσο πολλά, είναι νεκροί. Και ο κόσμος δεν ε, συγκλονίζεται ε, από το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Δεν καταλαβαίνει την κλίμακα της καταστροφής. Σου λέει ο κόσμος, ε, πλημμύρες συμβαίνουν συνέχεια, παντού στον κόσμο αλλά σιγά σιγά όταν άρχισαν τα πλάνα να έρχονται ε, όταν άρχισαν να έρχονται τα πλάνα λοιπόν στις τηλεοράσεις και τις δυτικές, κατάλαβε ο κόσμος ότι δεν ήταν άλλη μια πλημμύρα. Ήταν μια άνευ προηγουμένου θεομηνία αυτή η πλημμύρα. Και η διεθνής υποστήριξη ε, και η οικονομική σιγά σιγά άρχισαν να αυξάνονται. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση το εξωτερικό άρχισε σιγά σιγά να αυξάνεται και ελπίζουμε αύριο να είναι ακόμα μεγαλύτερη και θα έχουμε και μεγαλύτερε ε, επαφές και περισσότερε και συζήτηση για το πώς θα οικοδομηθεί υποστήριξη για την επόμενη φάση της ανοικοδόμησης. Και μετά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να κατανοηθούν. Ένα-δύο. Ε, υπάρχει μια κόπωση των δωρητών. Τέσσερις ήταν οι μεγάλες θεομηνίες, φέτος και μόνο. Ε, και η διεθνής προσοχή έχει στραφεί και προς τις άλλες θεομηνίες. Η Αιτία, ας πούμε, ήταν ε, τεράστια θεομηνία και ο κόσμος συνεισέφερε πάρα πολύ. Και ακολούθησαν οι πλημμύρες στο Πακιστάν. Δηλαδή, παρά την κόπωση αυτή των δωρητών, παρά τις θεομηνίες ε, που συμβαίνουν αρκετές και παρά την οικονομική κατάσταση στις Ηνωμένε Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα κράτη-μέλη σας ξέρετε ότι ε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Παρόλα αυτά, λέγω, η υποστήριξη που έχουμε είναι σημαντική και είμαστε ευγνώμονες και σας ευχαριστούμε γιατί πραγματικά μας δόθηκε βοήθεια και υποστήριξη. Και τέλος, για τη δημόσια συμμετοχή. Ναι, το ξέρω, το δέχομαι ότι θα πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερες εκστρατείες, να βγούμε προς τον κόσμο. Συμφωνώ απολύτως, αλλά θα ήθελα να σας πω και πάλι ότι έχουμε επιτυχίες. Και, ε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Γερμανία. Ο τηλεμαραθώνιος στη Γερμανία συγκέντρωσε χρήματα από τους Γερμανούς πολίτες και η ίδια η καγκελάριος προσωπικά πήγε στην τηλεόραση, στο στούντιο, κάθισε πάνω από 20 λεπτά για αυτό το σκοπό εκεί. Και πάνω από 218 εκατομμύρια ε, δολάρια συνέλεξε ο μέσος Γερμανός, ο Γερμανός πολίτης, έτσι, όχι η κυβέρνηση. Εδώ μιλώ για συνεισφορές των πολιτών, για τους ενάνους. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο υποθέτω ότι ε, εσείς εκπροσωπείτε ε, εκεί μια εκλογική περιφέρεια. Πάνω από 65 εκατομμύρια στερλίνες συνέλεξαν οι πολίτες στη Μεγάλη Βρετανία με τηλεμαραθώνιο, με ράνους, με διάφορες διοργανώσεις και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Στις 16 του μηνός ακολουθεί και άλλος μαραθώνιος έτσι, στο Λονδίνο. Μάλλον όχι, είναι ένα δείπνο ε, για συλλογή χρημάτων με τη διασπορά την πακιστανική στο Λονδίνο. Η Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και πάρα πολλοί άλλοι. Ε, που ζουν στην Ευρώπη, οι πολίτες των κρατών αυτών, ε, βοηθούν. Βεβαίως είναι πάντα ευπρόσδεκτα τα περισσότερα χρήματα, αλλά αναγνωρίζουμε τα όσα έχουν γίνει και είμαστε πρόθυμοι να βελτιώσουμε αν θέλετε και τη δική μας προσπάθεια για να συλλέξουμε περισσότερη βοήθεια. Θα ήθελα και πάλι να αναφερθώ τώρα σε δύο σημαντικές προσπάθειες που κάνουμε στο Πακιστάν και με τη διεθνή βοήθεια. Για τη διεθνή προσοχή και πώς αφυπνίσαμε τον κόσμο. Στις 19 Αυγούστου πήγα στον ΟΗΕ και μίλησα ε, ειδικά σε μια έκτακτη συνεδρίαση που είχε συγκληθεί για τις πλημμύρες. Και εκεί εκφράστηκε μεγάλη αλληλεγγύη προς το Πακιστάν. Και θαρρυντικό ήταν αυτό. Και μια δεύτερη τώρα εκδήλωση στις 19 Σεπτεμβρίου για μια δεύτερη πιο ενισχυμένη έκκληση του ΟΗΕ για 2 δις ε, δολάρια προς το Πακιστάν. Την πρώτη έκκληση που έκανε ο Γενικός Γραμματέας, πρέπει να σας πω ο κύριος Μπανκιμόν, 92% των ε, υποσχέσεων έγιναν πραγματικότητα, καταβλήθησαν τα χρήματα. Και δεν καθόλου εύκολο ε, υπό τις συνθήκες αυτές να δαπανηθούν τα χρήματα πραγματικά και να, και να δοθούν άλλο υποσχέσεις, άλλο η καταβολή των χρημάτων. Ε, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και αυτό. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να διδαχθούμε ε, από την ευρωπαϊκή εμπειρία. Έχει αναπτύξει ένα μοντέλο η Ευρώπη για πολλές περιφέρειες και η αν η Νοτιοανατολική Ασία προσπαθεί να δημιουργήσει μια κοινότητα σαν τη δική σας με τόση επιτυχία προσπαθεί να σας μιμηθεί και στη Νότια επίσης Ασία ε, πρέπει να διδαχθούμε και εμείς από εσάς και από το παράδειγμά σας. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό στην Νότια Ασία και τη περιφέρεια στην οποία αναφέρεστε, πρέπει οι Ευρωπαίοι να βοηθούν και να υποστηρίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις δημοκρατικές κυβερνήσεις. Γιατί οι πολιτικοί και οι δημοκράτες εν γέννη προσπαθούν να λύνουν τα ζητήματα μέσω διαλόγου και όχι μέσω των πολέμων. Αυτό μας διδάσκει και η ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν διαθέσιμοι να το κάνουν. Το ΣΑΡΚ είναι μια πολύ ε, καλή ευκαιρία. Δεν χρησιμοποιείται ε, όσο θα έπρεπε αυτή η δυνατότητα, αυτό το φόρουμ. Και το αναγνωρίζω στο Μπουτάν, στον την τελευταία φορά που ε, συνεδριάσαμε, ε, μας προβλημάτισε αυτό. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την περιφερειακή συνεργασία, πώς μπορούμε να κάνουμε πιο αποδοτικές τις συνεδριάσεις. Θα βελτιωθούμε, είμαι βέβαιος θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα σας φτάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αρλάκη, παρακαλώ, που είναι συγγητής μας για το Αφγανιστάν και μόλις προηγουμένως συζητούσαμε ορισμένες από τις τροπολογίες της εκθέσεώς του πριν έρθετε εσείς. Έχετε το λόγο, παρακαλώ, κύριε Αρλάκη. Ναι, δύο σύντομες ερωτήσεις, ε, κύριε Υπουργέ. Η μία αφορά την ε, περιφερειακή λύση του αφγανικού προβλήματος και το άλλο αφορά τα ναρκωτικά στο Αφγανιστάν. 27 χώρες ε, βρίσκονται τώρα στο αφγανικό έδαφος για κάποιο είδος παρέμβαση και ορισμένες από αυτές δεν παρεμβαίνουν και κατηγορούν ότι το Πακιστάν ότι παρεμβαίνει εκεί στο Αφγανιστάν. Είναι, κάποιο, είναι κάπως παράδοξο και με έχει πολλές φορές απασχολήσει να βλέπω διαμαρτυρίες για το ότι αναμειχνείται το Πακιστάν. Η χώρα μου είναι 2.000 ε, χιλιόμετρα μακριά και αναμειγνύεται. Εσείς που είστε, ε, έχετε κοινέ, κοινά σύνορα, λαό, γλώσσα, ποια είναι η παρέμβαση των περιφερειακών δυνάμεων στο Πακιστάν. Ποια είναι η περιφερειακή λύση για το αφγανικό πρόβλημα κατά την άποψή σας, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να είναι μια μεγάλη συνεισφορά, συμβολή. Και δεύτερον, πώς βλέπετε το θέμα των ναρκωτικών. Το Πακιστάν είναι ένα από τα μεγάλα θύματα μαζί με το Ιράν σε περιφερειακή κλίμακα όσον αφορά την παραγωγή οποίου το Αφγανιστάν και γιατί οι ευρωπαϊκές προσπάθειες οι προσπάθειες της διεθνού κοινότητας για την ε, κρίζωση του σκαλέριας το οποίο απέτυχαν τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η κυρία Μπόσκουρτ τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την εισήγησή σας ε, που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν να σας πω ότι όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο Παρακολουθούμε την κατάσταση με τις πλημμύρες με μεγάλη ε, ανησυχία και επίσης με, μεγάλη συμπάθεια συζητήσαμε πριν από λίγες εβδομάδες για το θέμα της, ε, των συμφωνιών επανεισδαχής λόγω του προβλήματος με τις, με τις πλημμύρες. Τι θα γίνει ο κόσμος. Θα τους στέλνουμε στο Πακιστάν όταν η ίδια η χώρα έχει τεράστια προβλήματα με μετατοπισμένους πληθυσμούς. Το ίδιο θέμα για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το θέμα της Σύμβασης της Γενέβης για τους πρόσφυγες, που δεν έχει υπογραφεί από το Πακιστάν. Τώρα άκουσα να λέτε στην εισήγησή σας ότι το Πακιστάν υπέγραψε σήμερα ε, όλες τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή αυτό σημαίνει πως την υπογράψατε τη Σύμβαση της Γενέβης. Ή ότι είναι σχεδιασμένη η υπογραφή. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση αφορά το εξή. Εσεί ε, αναφερθήκατε σε πολλά σημαντικά θέματα, αλλά όχι στην κατάσταση των γυναικών στο Πακιστάν, που είναι πολύ σημαντικό θέμα για μένα. Μιλήσατε για τον αγώνα κατά τις στόχες αλλά η εκπαίδευση των γυναικών είναι ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα κατά της στόχια. Όταν κανείς εκπαιδεύσει τις γυναίκες θα εκπαιδεύσει μια ολόκληρη οικογένεια ταυτόχρονα, πράγμα που θα ε, οδηγήσει σε πρόοδο ολόκληρη την κοινωνία. Το ίδιο σημαίνει και για την ε, συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία της χώρας. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια περισσότερο για την κατάσταση και για το ποια είναι τα σχέδια του της κυβέρνησης για τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ. Υπουργέ. Είστε εξαιρετικά διπλωματικός και εγώ είμαι και διπλωματικός στην ε, βασική μου εκπαίδευση, αλλά τώρα κάνω την πολιτικό, άρα θα τα πω ομά. Νομίζω ότι έχουμε ένα μεγάλο δίλημα στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη σε σχέση με το Πακιστάν, διότι ναι, βλέπουμε την ανάγκη στον... του να βοηθήσουμε το Πακιστάν. Αλλά πιστεύουμε επίσης ότι το Πακιστάν έχει τεράστιες δυσκολίες να αυτοβοηθηθεί. Και αυτό έχει να κάνει με τη φύση της διακυβέρνησης. Αν δηλαδή πρόκειται για πραγματική δημοκρατία ή όχι. Ή αν είναι μόνο κατόνομα δημοκρατία. Ο φόβος είναι Μήπω όλη ε, η κυβέρνηση δεν, είναι, δεν έχει τον έλεγχο. Αυτός που έχει τον έλεγχο μήπω είναι ο στρατό και η ε, στρατική αντισκατοσκοπία. Και γι' αυτό βλέπουμε τόσα πολλά προβλήματα. Και φυσικά και στι σχέσει με την Ιδία, εγώ πρώτη και καλύτερη συμφωνώ πω το Κασμίρ είναι διεθνέ ζήτημα και ότι χρειάζεται διεθνή ε, παρέμβαση για να λυθεί το πρόβλημα του Κασμίρ. Μα, αλλά το Πακιστάν δεν έχει βοηθήσει ώστε να ε, δοθεί αυτή η διεθνής ε, βοήθεια να υπάρξει αυτή η διεθνής ανάμειξη ιδιαίτερα λόγω του ρόλου που παίζουν αυτοί που υποστηρίζουν την τρομοκρατία κατά της Ινδίας. Και φυσικά και εγώ ναι, αναθέτω πολλές ελπίδες στο δημοκρατικό διάλογο με την Ινδία. Αλλά αυτό δεν μπορεί να σταθεί αν ταυτόχρονα συνεχίζονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Ινδίας όπως στη Βομβάη και ούτω καθεξής και το ίδιο ισχύει και με το Αφγανιστάν. Βεβαίως, εκτός από τις σχέσεις που είπε ο συνάδελφο Αρλάκη ότι ναι, έχετε σύνορα κοινά, ότι έχετε κοινό, κοινά στοιχεία με ίδιο λαοί κτλ. Και πάλι βλέπουμε πολλέ φορές ότι παρεμβαίνεται, υπάρχει παρέμβαση. Και φυσικά υπάρχει πακιστανική παρέμβαση και αυτή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, αλλά πιο συχνά είναι αρνητική. Και την έχω δει αυτή την παρέμβαση το 97-98 όταν ο πρέσβης του Πακιστάν στον ΟΗΕ έφερνε μαζί του τον εκπρόσωπο του καθεστώτος των Ταλιμπάν για να καθίσει στη θέση του Αφγανιστάν και να αρχίσει να πιέζει τους, ε, τους ε, υπόλοιπους διπλωμάτες. Η παρέμβαση λοιπόν υπάρχει. Θετική ή αρνητική. Φοβούμαι όμως πως είναι πιο αρνητική αν δεν είναι η δημοκρατική κυβέρνηση που ελέγχει τα πράγματα και εξακολουθεί να είναι το ISI. Για μένα η ενδοπακιστανική σύγκρουση για το Κασμίρ είναι ίσως το πιο επικίνδυνο πρόβλημα για την παγκόσμια ασφάλεια. Όχι μόνο για την ασφάλεια του Πακιστάν και της Ινδίας, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, γιατί μιλάμε για δύο πυρηνικές δυνάμεις. Και τι γίνεται με το NPT, με τις τελευταίες εξελίξεις και την τελευταία διάσκεψη του NPT, όταν ο πρόεδρος Ομπάμα μιλά για έναν, άνθρωπο, έναν κόσμο ελεύθερο από πυρηνικά, απαλλαγμένο από τα πυρηνικά όπλα. Εσείς τι λέτε. Και να αναφέρω επίσης και υποστηρίζω τα όσα είπε η συνάδελφος Βοσκούρτ για το θέμα του ρόλου της παιδείας των γυναικών. Μια δημοκρατική κοινωνία χρειάζεται να εκπαιδεύσει τις γυναίκες. Όντως είναι ο τρόπος για την καταπολέμηση της στόχης. Στο Πακιστάν υπάρχουν φοβερά προβλήματα, εγκλήματα, βία κατά των γυναικών. Τι κάνει η κυβέρνησή σας για όλα αυτά. Και αυτό έχει επίσης να κάνει με το πρόβλημα της παιδικής εργασίας θέματα τα οποία θα προκύψουν με τη συμφωνία για περισσότερες εξαγωγές ε, από το Πακιστάν. Είναι ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά είναι και θεμητός ανταγωνισμός, δίκαιος ανταγωνισμός. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα να σας ρωτήσω δεν μπορούσα να είμαι εδώ στην συζήτηση για το Αφγανιστάν, γιατί ήμουν σε μια άλλη συνεδρία όπου συζητούσαμε κατά της θανατικής ποινή. και μόλις έμαθα ότι το Πακιστάν έχει περίπου 7.500 ανθρώπους που είναι καταδικασμένοι σε θάνατο. Αν και δεν εκτελεί τις ποινές, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στο Πακιστάν, στον κόσμο και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, μάλιστα, ανάμεσα στους καταδικασμένους σε θάνατο με ευρωπαϊκή υπηκότητα. Και το Πακιστάν ξέρω πως έχει μια πολύ, ένα πολύ ικανό και ζωντανό δικαστικό σώμα. Πώς μπορεί λοιπόν η δημοκρατική κυβέρνηση του Πακιστάν να σημάνει διαφορά και να χειριστεί αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινήσω από εσά. Μιλήσατε για το Αφγανιστάν και την ανάμεξη του Πακιστάν στο Αφγανιστάν. Φαντάζομαι ότι μιλάτε για ανάμεξη, μιλάτε για αρνητική ε, παρέμβαση. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό μπορεί να ίσχυε στο παρελθόν, αλλά τα πράγματα επί τόπου έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό σήμερα. Σήμερα, μην ρωτάτε εμένα, ρωτήστε τον Υπουργό Εξωτερικών του Αφγανιστάν, το Πρόεδρο του Αφγανιστάν, ή βουλευτές του Αφγανιστάν. Και νομίζω είμαι πεπισμένος πως η άποψή του σήμερα θα είναι διαφορετική. Σήμερα το Πακιστάν και το Αφγανιστάν έχουν ένα διαφορετικό είδος σχέσης που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και βελτιώνεται διαρκώς. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Ναι, 2.500 χιλιόμετρα είναι τα κοινά μας σύνορα. Πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς τόσα σύνορα. Αλλά ποτέ στο παρελθόν, από τότε που δημιουργήθηκε η χώρα, δεν έχουμε αναπτύξει τόσα στατεύματα για τη διαχείριση μόνο των σύνορων. 150.000 άνθρωποι είναι στα σύνορα. Ποτέ α, πριν δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Σχεδόν χίλιοι συνοριακοί σταθμοί έχουν δημιουργηθεί σε όλα τα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν για να βελτιωθεί η διαχείριση των σύνορων. Έχουμε μια επιτροπή που συντονίζει τα συνοριακά θέματα για τον Αφγανικό στρατό, ISAF και Πακιστανικό στρατό. ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση αυτών των συνόρων. Η εισαγωγή επίσης νέα τεχνολογίας έχει γίνει, βιομετρικά συστήματα και ούτω καθεξής, ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση των συνόρων στο Αφγανιστάν, ε, με το Αφγανιστάν. Έγιναν προεδρικέ εκλογές στο Αφγανιστάν. Για πρώτη φορά ο πρόεδρο Καρζάη και πολλοί από του συναδέλφου του, καθώ και ο υποψήφιο που έχασε τι εκλογέ από τον Υπουργό Εξωτερικών, Αμπτούλα Αμπτούλα. Αναγνώρισαν δημόσια πως το Πακιστάν δεν είχε κανέναν ε, δικό του υποψήφιο. Δεν αναμίχθηκε. Εμείς είπαμε ότι ο λαός του Αφγανιστάν πρέπει να επιλέξει ποιον θέλει για να τον κυβερνήσει. Εμείς πρέπει να συνεργαστούμε με την Καμπούλ. Πρέπει να ρυθμίσουμε τις σχέσεις μας με την Καμπούλ. Παλιότερα το Πακιστάν καθοριζόταν από μία εθνοτική ομάδα, τους Παστούν, και ξέρετε ότι οι Ταλιμπάνοι περισσότεροι προέρχονται από αυτή την φυλή. Εμείς τώρα συνομιλούμε με άλλες φυλές, με τους Φαζάρα και άλλους που είναι, ε, ήταν πέρα από τις επαφές και αυτό αναγνωρίζεται από τους Αφγανούς, από τους ανθρώπους που αυτοί διαμαρτύρονταν για αυτά τα θέματα. Σήμερα αναγνωρίζουν πώς τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που εξελέγει η δημοκρατική κυβέρνηση για τα ναρκωτικά. Να σας πω ότι σήμερα το Πακιστάν δεν έχουμε, έχουμε μηδέν καλλιέργεια παπαρούνας. Τα καταφέραμε. Εκριζώσαμε τις παπαρούνες. Αλλά το θέμα του Αφγανιστάν, τα ναρκωτικά στο Αφγανιστάν είναι σημαντικό θέμα. Και το έχουμε συζητήσει, το έχουμε θίξει και στη συνεδρίαση στο Παρίσι και μου είπαν ότι δεν ήταν τμήμα της εντολής του ΝΑΤΟ και ρώτησα τότε τότε να διευρύνετε την εντολή σας, να το βάλετε στην εντολή σας, γιατί τα λεφτά των ναρκωτικών χρησιμοποιούνται από το στρατό, από τους ταραξίες και είναι ένας ε, από τους πόρους που έχουν. Και πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε θετικά και να έχουμε μια πιο περιφερειακή προσέγγιση σε αυτό. Εσείς είπατε τι γίνεται με τις περιφερειακές λύσεις. Ναι, το Πακιστάν σήμερα έχει αναγνωρίσει και υποστηρίζει περιφερειακή λύση. Σήμερα είμαστε σε διάφορες διαδικασίες, προσπαθούμε σε τριμερείς διαδικασίες που προωθούν την περιφερειακή ανάμειξη με το Ιράν. Και το Ιράν συνορεύει και με το Πακιστάν και με το Αφγανιστάν. Πώς μπορούμε να γνωρούμε το Ιράν λοιπόν όταν μιλάμε για σταθερότητα και ειρήνη στο Αφγανιστάν. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Συνεργασία ανάμεσα στις τρεις χώρες. Από την άλλη μεριά έχουμε το Τατζικιστάν, άλλος σημαντικός ε, γείτονας. Προσπαθούμε να κάνουμε πάλι και εκεί τριμερή συνεργασία. Άλλη τριμερή συνεργασία με τη ΣΥΠΑ. Αφγανιστάν, Πακιστάν, είπα. Ή ε, και πολυμερή συνεργασία ανάμεσα Τατζικιστάν, Αφγανιστάν, Πακιστάν και Ρωσία. Η ε, Ρωσία έχει μεγάλη επιρροή στις ε, κεντρικές εκεί δημοκρατίες. Είναι ένας παγκόσμιος παίκτη. Και έχει πολύ ισχυρή τοπική περιφερειακή παρουσία και με αυτούς πρέπει να κάνουμε χωριό. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μια περιφερειακή λύση για το Αφγανιστάν και συμφωνούμε με αυτό που είπατε ότι αυτή είναι η μακροπρόθεσμη λύση για το Αφγανιστάν. Τώρα, κάτι που εσείς είπατε σε σχέση με το Αφγανιστάν. Ότι εμείς ε, είχαμε επαφές με τους Ταλιμπάν και ότι εκπρόσωπος των Ταλιμπάν ε, στην ουσία... Νομίζω εσείς το είπατε. Α, ναι, εσείς το είπατε, κύριε μου. Ότι το επιτράπηκε να καθίσει στον ΟΙΕ, εν περιπτώσει, σε κάποια αίθουσα. Μα αυτά έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει. Σήμερα στο Πακιστάν έχουμε καταλάβει ότι δεν θέλουμε να ταλιμπανοποιηθούμε. Άμα δεν θέλουμε να τα λιμπανοποιηθούμε, λοιπόν, το πρώτο και κύριο που πρέπει να κάνουμε είναι να μην τα λιμπανοποιηθεί και το Αφγανιστάν. Άμα κερδίσουν έδαφο οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, θα είμαστε οι επόμενοι. Σήμερα έχουμε ανθρώπους στην κυβέρνηση που είναι κατά αυτού του είδους σκέψης, αυτών των αρχών. Ο κόσμος λοιπόν που είναι τώρα στην εξουσία στο Πακιστάν είναι κόσμος που μπορεί να καταλάβει αυτά που λέτε, μπορεί να καταλάβει τις ανησυχίες σας και μπορεί να έχει επαφή μαζί σας και να φτιάξει εταιρικέ σχέσεις μαζί σας. Σήμερα στο Πακιστάν έχουμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι φίλη και, και συνεταίρη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ρωτήσατε επίσης ποιος ελέγχει την κατάσταση η στρατιωτική, η ΆΙΣΑΠ. Ξέρετε ότι έχουμε, ε, είχαμε πολλές στρατιωτικές κυβερνήσεις και στρατιωτικές ε, παρεμβάσεις τις τελευταίες έξι δεκαετίες. Αυτό είναι αλήθεια. Και εμείς ως δημοκράτες ε, στο κόμμα το οποίο εγώ αντιπροσωπεύω είμαστε το κόμμα το οποίο συστηματικά ήταν αντίθετο με το στρατιωτικό νόμο στο Πακιστάν, ήταν ο Ζέο, ο Γιούμπ ή ο οποιοδήποτε. Δυστυχώς δεν ακουστήκαμε. Οι Βρυξέλλες δεν μας πρόσεχαν όταν δεν ήμασταν στην κυβέρνηση, ούτε η Ουάσιγκτον μας άκουγε. Τότε έπρεπε να στηρίξετε κόσμο σαν και που λέγανε Στηρίξτε τα δημοκρατικά, τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ε, ε, στηρίξτε την ηγεσία που είναι σε, στην εξορία. Δώστε μας τη φωνή που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια δημοκρατική κουλτούρα, νοοτροπία στο, στο Πακιστάν. Ευτυχώς αυτό έγινε πραγματικότητα πια και οι, δημο, οι Ευρωπαίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Είμαστε ευγνώμονες, στείλατε παρατηρητές, εμείς φοβόμασταν. Δεν ξέραμε καν αν θα γίνονταν ε, ελεύθερα οι εκλογές φέτος. Με τη δική σας παρέμβαση και το δικό σας ενδιαφέρον το πετύχαμε. Και γι' αυτό είμαι και σήμερα εδώ. Με χωρίς τη βοήθειά σας δεν θα ήμουνα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν γι' αυτό αλλά πρέπει βέβαια να συνεχίσουμε για με το πέρασμα του χρόνου καθώς θα ριζώνει η δημοκρατία και η πολιτική ηγεσία θα επιβεβαιώνεται ακόμα περισσότερο, θα αισθάνεται πιο σίγουροι. Είμαστε βέβαιοι ότι πρέπει ο στρατός να παίξει το ρόλο του που είναι ο συνταγματικός ρόλος του στρατού. Αλλά όχι στη διακυβέρνηση. Η διακυβέρνηση ανήκει στους εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού μέσω των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών κάθε πέντε χρόνια που είναι ο χρόνος θητείας του Κοινοβουλίου μας. Και πάλι είμαστε συνεταίροι, συνεταίροι στην να αναπτυχθούμε περισσότερο, να ενισχύσουμε και να ενισχυθούμε, να ενισχύσουμε τη φωνή μας και να εξασφαλίσουμε τους θεσμούς μας στην μια γραμμή πολιτικής ε, ηγεσίας. Να σας πω και να σας διαβεβαιώσω ότι σήμερα, για να είμαστε δίκαιοι, έχουμε επικεφαλή στο στρατό έναν άνθρωπο ο οποίος ανέκαθεν ήταν ε, δημοκρατικός. Και μάλιστα διευκόλυνε τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Και ακολουθεί τη γραμμή και στηρίζει την εκλεγμένη κυβέρνηση. Φυσικά παίρνει χρόνο η αλλαγή ώστε να δημιουργηθεί μια νοοτροπία η οποία δεν έχει αναπτυχθεί εδώ και δεκαετίες. Και ο κόσμος χρηματοδοτούσε και συνεργαζόταν με αυτούς εκεί. Ε, αυτό θα πάρει χρόνο. Οι παλιές συνήθειες αργά-αργά ε, ε, ξεριζώνονται. Είμαστε σε μια διαδικασία μεταβατική και με το πέρασμα του χρόνου θα ριζώσει, θα ριζώσει και θα δυναμώσει. Πρέπει να επιμείνουμε και να είμαστε υπομονετικοί. Αλλά θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε, είμαι βέβαιος. Να μιλήσω και για τις γυναίκες. Να σας πω σήμερα πως έχουμε ε, πολλές μορφωμένες καλλιεργημένες γυναίκες. Μία από αυτές είναι εκεί, η γερουσιαστής ε, Ζαϊνάμπ Αμάρ. Και όταν προετοιμαζόμασταν για τη συνάντηση στι Βρυξέλλε, τη ζήτησαν να έρθει και να κάνει μια από τι εισηγήσει. Γιατί, για να δει ο κόσμο ότι έχουμε γυναίκε βουλευτίνε που έχουν δικό τους λόγο Σήμερα οι γυναίκες παίζουν έναν πιο ε, ε, σημαντικό ρόλο. Λάτε να δείτε το κίνημα των δικηγόρων, των νομικών, πώς οι γυναίκες νομικοί του Πακιστάν παίζουν εξέχοντα ρόλο. Ελάτε να δείτε τις ΜΚΟ που τις ε, δικούν οι γυναίκες με ικανότατο τρόπο. Επίσης, πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι στο Πακιστάν είναι γυναίκες και παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο δικαστίνες αρχιτεκτόνησες, μηχανικοί, διπλωμάτες, αντιπροσωπεύουν το Πακιστάν σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και είμαστε γιατί, περήφανοι για αυτές γιατί παίζουν εξαιρετικό ρόλο. Η Μπεναζίρ Μπούτο έδωσε το φως, αντιστάθηκε σε μια δικτατορία όταν κανείς δεν την έδινε σημασία και δεν την άκουγε. Αλλά αυτή επέμεινε. Συνέχισε. Και μέχρι και τη ζωή της. Υπάρχουν παραδείγματα, όπως τα αναφέρατε. Κακά παραδείγματα, αλλά είναι μειονότητα. Μειοψηφία. Ακόμα και η Ισλαμική κουλτούρα δεν επιτρέπει αυτά, αυτές τις ακρότητες. Αυτά είναι αρχαϊκά τα έθιμα. Η θρησκεία μας δεν τα επιτρέπει, η νομοθεσία μας δεν τα επιτρέπει, ούτε το σύνταγμά μας τα επιτρέπει. Και γι' αυτό λοιπόν, λοιπόν συμφωνούμε μαζί σας. Το πυρηνικό θέμα. Ζήτημα. Ναι, είμαστε σήμερα πυρηνική δύναμη αλλά έχει τελείω αμυντική φύση. Δεν, έχουμε, δεν θέλουμε να επεκταθούμε. Απλώ ε, είναι ένας μηχανισμός αμυντικό. Σε αντίδραση στη χώρα τη γειτονική που προχώρησε γνωρίζοντας το μέγεθος και την έλλειψη ισορροπίας που έχουμε μεταξύ μας έπρεπε να το κάνουμε κι εμείς. Ευτυχώς όμως σήμερα με τον γείτονα χώρα μας Έχουμε μαζί βρει από κοινού πυρηνικές συμφωνίες. Και παρά τις εντάσεις και παρά τις δυσκολίες έχουμε τιμήσει τις συμφωνίες αυτές γιατί και δύο πλευρές αναγνωρίζουμε και συνειδητοποιούμε πόσο λεπτό είναι αυτό το θέμα και πόσο ασφαλισμένα θα πρέπει να είναι όλα αυτά τα συστήματα. Και όταν μιλήσατε για την ε, διάσκεψη κορυφής του Ομπάμα στη Ουάσιγκτον, ναι, προσκεκλήθη το Πακιστάν και συμμετείχε. Και υπήρχε ομοφωνία εκεί πέρα, ότι η ειδική αρχή και τα συστήματα ασφαλείας που έχουμε είναι τόσο ασφαλή όσο και οποιοδήποτε άλλο νου. Οπότε αυτό αναγνωρίζεται. Και δεν ε, παραβλέπουμε τις ανησυχίες σας. Τώρα, εσείς μιλήσατε για ανθρώπινα δικαιώματα. Πάντοτε υπάρχει χώρος για βελτίωση σε αυτούς τους τομείς και εδώ έρχεται μια επίσημη κυβέρνηση που είναι ευαίσθητη στα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε είναι τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των γυναικών. Μιλήσατε για παιδική εργασία, μιλήσατε για άλλα θέματα, μιλήσατε και για τη θανατική ποινή. Ναι, γίνεται η συζήτηση, γίνεται η συζήτηση. στη χώρα για το αν θα πρέπει να σε διατηρηθεί ή όχι. Υπάρχουν χώρες που ισχύει Κάποιες πολιτείες της είπα, πολλές, έχουν ακόμα τη θενατική ποινή. Υπάρχει ο κόσμος που είναι αντίθετος, γίνεται η συζήτηση όπως σας είπα. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά έχουμε νομικούς. Οι 7.500 που αναφέρατε αντιπροσωπεύονται. Υπάρχουν δικηγόροι που τους υποστηρίζουν και τους αντιπροσωπεύουν. Ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε λάβει μέτρα για να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ε, συμμορφωθούμε προς τα διεθνή στάνταρ. Αναφέρατε τους πρόσφυγες. Νομίζω ότι έχει αναγνωριστεί ότι Ακόμα και σήμερα έχουμε σχεδόν 3 εκατομμύρια πρόσφυγες στο Πακιστάν και είναι όλοι αυγανοί πρόσφυγες. Έχει αναγνωριστεί παγκοσμίω. Ο κόσμος τους ξεχνά, αλλά εμείς τους προσέχουμε, τους στηρίζουμε. Ακόμα και σήμερα πάνω από 150.000 φοιτητέ, αυγανοί φοιτητέ, από, από αυτά τα στρατόπεδα προσφύγων συμμετέχουν στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. 6.000 φοιτητέ Πολλοί από αυτά τα στρατόπεδα προσφύγων από τις προσφυγικές οικογένειες φοιτούν στα διάφορα μας ε, ε, πανεπιστήμια στο Πακιστάν. Δεδομένου των πόρων, νομίζω πως δεν τα καταφέρνουμε κάσχημα. Επίσης μιλήσατε για το θέμα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Βομβάη. Σήμερα, ε, συγγνώμη, εκείνη την ημέρα βρισκόμουν στο Δελχή όταν έγινε αυτό, ε, αυτή η φρικτή τρομοκρατική επίθεση. Τι έκανα εκεί. Προσπαθούσα να φτιάξω γέφυρες, να δημιουργήσω, να, να συνεννοηθώ, να τους ζητήσω να προχωρήσουμε στα θέματά μας. Έγινε η επίθεση. Τώρα. Η αντίδραση σε αυτή την υπόθεση δεν έπρεπε να είναι πάυση των διαπραγματεύσεων όπως ήταν η άμεση αντίδραση των Ινδών. Η αντίδραση σε αυτό θα έπρεπε να είναι περισσότερη συνεργασία. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί η τρομοκρατία δεν αφορά πια συγκεκριμένες χώρες. Δεν είναι ότι η Ινδία χτυπήθηκε από τους τρομοκράτες. Πολλά άλλα κράτη της περιοχής έχουν χτυπηθεί από την τρομοκρατία και τους τρομοκράτες και εμείς οι ίδιοι υποφέρουμε από αυτό. Εμείς είχαμε περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Πακιστάν τα τελευταία χρόνια από ό,τι μπορούν ποτέ να φανταστούν οι Ινδοί. Αυτό τι σημαίνει. Σήμερα η κοινή γνώμη στο Πακιστάν είναι και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις αρνητικές επιπτώσεις της τρομοκρατίας, τις οικονομικές επιπτώσεις της τρομοκρατίας, τις κοινωνικές και τις πολιτικές επιπτώσεις της τρομοκρατίας. Δηλαδή, <coughs> είμαστε πιο έτοιμοι να δουλέψουμε μαζί τους και σκοπεύουμε να το κάνουμε. Είναι ένας κοινό εχθρός. Κοινό εχθρός και χρειάζεται κοινή προσέγγιση για να τον αντιμετωπίσουμε. Για το Κασμίρ είπα ότι είναι ένα θέμα το οποίο αναγνωρίζετε και εσείς οι ίδια το είπατε ότι το αναγνωρίζετε ως διεθνές ζήτημα, διεθνής ε, δια... διαφορά. Υπάρχουν διεθνείς δεσμεύσεις σε ψηφίσματα του, του, του ΟΗΕ. Υπάρχει τρόπος να προχωρήσουμε και να το λύσουμε με ειρηνικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ εξοχότατε. Νομίζω ότι ήταν μια καλή ευκαιρία αυτή να συζητήσουμε. Έχουμε πολλά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ελπίζω να είστε ικανοποιημένος. Εγώ είμαι και εξ ονόματος της Επιτροπής μου, πρέπει να σας το πω. Γνωρίζετε ε, ότι είναι και ελπίζω να είναι ικανοποιημένοι και οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ εξοχότατε και εσάς και την αντιπροσωπεία σας για τη συνεδρίαση αυτή. Καλή σας επιτυχία. Έχετε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσετε. Ελπίζω τελικά όμως να φτάσουν όλα σε αίσιο πέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη. I would like to, we uh, leave, I would like... Πριν φύγουμε, θέλω να ενημερώσω τους συναδελφούς ότι στις 18 του μηνό στο Στρασβούργο, 7 με 9 το βράδυ, τη Δευτέρα, θα ψηφίσουμε για το βραβείο Σαχάροφ. Ενώ στις 19 του μηνός, 5 μέχρι το απόγευμα, θα συνεδριάσουμε, θα δεχθούμε στη συνεδρίαση αυτή τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Μπαν Κιμούν, για να το γνωρίζετε αυτό.